Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σε όλους. Με χαρά καλωσορίζω εκ μέρους ε, της ε, Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας τον κύριο Μπίλιτσα, που είναι ειδικό απεσταλμένος για τον αφοπλισμό και την μη διάδοση επικεφαλής της διεύθυνσης ΣΕΚΠΟΛ 1 για τον αφοπλισμό, μη διάδοση και έλεγχο των εξαγωγών όπλων, τον κύριο Βίλιαμ Αλμπέρκ, διευθυντή του Κέντρου Ελέγχου Εξοπλισμών, Αφοπλισμού και Μη Διάδοση Όπλων μαζική καταστροφή του ΝΑΤΟ και τον κύριο Μπρούνο Λετέ, αναλυτή για το German Marshall Fund ε, των ΗΠΑ. Στι 2 Αυγούστου το καλοκαίρι φέτο, η διεθνή κοινότητα διαπίστωσε ότι κατέρευσε η συνθήκη INF ε, για την εξάλληψη των ε, ε, μέσου ελληνικού. που ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμια, του παγκόσμιου συστήματος για το, τον έλεγχο των εξοπλισμών και συνεισέφερε επί τρει δεκαετίε και παραπάνω στην ειρήνη και σταθερότητα για τα πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Φεβρουάριο, ε, λίγο πριν ε, ανακοινωθεί από τη Ρωσία και τι ΗΠΑ η πρόθεσή του να αναστείλουν την υποχρέωσή του με βάση τη, τη συνθήκη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε ένα ψήφισμα για το μέλλον τη συνθήκη INF και την επίπτωσή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το ψήφισμα τονίζαμε ότι η κατάρρευση της συνθήκης θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την ασφάλεια στην Ευρώπη. Το τέλος της συνθήκης ΑΕΝΕΦ ε, θέτει σημαντικές απειλές σε παγκόσμιο επίπεδο και κατά πάσα πιθανότητα θα θέσει σε κίνδυνο τη διαδικασία επέκτασης και άλλης μιας σημαντικής συνθήκης, τη συνθήκης New Start. Αν η New Start δεν παραταθεί πριν από το Φεβρουάριο του 2021, ο πλανήτη μα δεν θα έχει πλέον κανένα περιορισμό που θα είναι νομικά δεσμευτικό για του πυρηνικού εξοπλισμού. Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια λοιπόν μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο. και θέλουμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίζει όλο και περισσότερο ενεργό ρόλο και να ξεκινήσει διαπραγματεύσει για μια πολυμερή συμφωνία για τον έλεγχο των εξοπλισμών. Και θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Μπίλτσα να μας μιλήσει για τη δική του άποψη για το μέλλον του καθεστώτος της μη διάδοσης και για τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε η, ο πολυμερής πυρηνικός αφοπλισμός να είναι ένα από τα θέματα που αποτελούν προτεραιότητα στο θεματολόγιο ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους επόμενους ομιλητές. Είναι το λόγο στον κύριο Μπίλτσα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ για την εκλογή σας ως πρόεδρος αυτής της Επιτροπής που είναι βασική επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλω να σας διαβεβαιώσω για την πλήρη στήριξη και για τη συνεργασία των δομών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που ασχολούνται με τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση και τον έλεγχο εξαγωγών όπλων. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην Επιτροπή σας. Έχω την τιμή να παρευρίσκομαι σε αυτό το βήμα με διακεκριμένους εμπειρογνώμονες και συναδέλφους από το Γενικό Επιτελείο του ΝΑΤΟ και από τη γενικότερη κοινότητα των ερευνητών. Φοβούμαι ότι ε, είναι συμβολικός ο χαρακτήρας του ότι μια από τις πρώτες συζητήσεις ε, για τη νέα θητεία της, Επιτροπής, της Υποεπιτροπής ΣΕΝΤΕ ασχολείται με τα θέματα αυτά. Η μη διάδοση, ο αφοπλισμός, ο έλεγχος των όπλων και των εξαγωγών όπλων αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την πολιτική ασφάλεια. Η συνθήκη INF ήταν ένα βασικό θέμα των συζητήσεων της Επιτροπής ΣΕΝΤΕ στο παρελθόν, ιδίως στις 23 Ιανουαρίου του 2019 και το αποτέλεσμα ήταν και ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Φεβρουαρίου του 2019. Θέλω να σας δώσω κάποια γενικά στοιχεία για το υπόβαθρο. Κάθε φορά που ακούω να περιγράφεται η συνθήκη INF ως μια ρύθμιση για τον έλεγχο των όπλων της εποχής του ψυχρού πολέμου ε, μου φαίνεται πολύ περίεργο και δεν συμφωνώ καθόλου, γιατί δεν είναι, ε, δεν είναι πρόκειτο περί αυτού. Καταρχήν, ήταν ένα από τα βασικά έγγραφα που βοήθησαν να λήξει ο ψυχρός πόλεμος και πιο σημαντικά μας βοήθησε για την εξάλληψη μιας μεγάλης κατηγορίας όπλων, ε, πυράβλων και εκτοξευτήρων, συνεισφέροντας στον αφοπλισμό, όχι μόνο στον έλεγχο των εξοπλισμών. Τα βασικά γεγονότα ήταν ότι η συνθήκη για την εξάλληψη των πυράβλων μέσου και βραχύτερου βεληνικού ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευση μεταξύ ΗΠΑ και ε, Σοβιετική Ένωση, μεταξύ Ρίγκαν και Γκορμπατσόφ, ε, στη διάσκεψη κορυφή του Ρέκεβικ το 1986 και υπεγράφει το 1987 και τέθησε ισχύ το 1988 ανέλαβαν την ευθύνη οι δύο χώρες να καταστρέψουν ε, το ε, ε, τους εκτοξευόμενους από έδαφο βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους κρούς με πελληνικές 500 5.500 χιλιόμετρα καθώς και τους εκτοξευτές τέτοιων πυράβλων. Μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Λευκορωσία, το Καζακστάν και η Ουκρανία ήταν οι χώρες διάδοχοι που έγιναν μέρη της INF. Παρόμοιες απαγορεύσεις δεν ίσχυαν για την Κίνα και άλλες χώρες της Ασίας. Τον Ιανουάριο του 2007 ο πρόεδρο ε, Πούτιν δήλωσε ότι η συνθήκη INF δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα ασφάλεια τη Ρωσία πλέον και παρόμοιε δηλώσει ακολούθησαν και από του στρατιωτικού τη Ρωσία. Από το 2014 οι Ηνωμένε Πολιτείε άρχισαν να κατηγορούν δημοσίω τη Ρωσία ότι παραβιάζει τι ε, υποχρεώσει τη συνθήκη INF. Η Ρωσία το αρνήθηκε και έκανε αντίστοιχε αντίθετε κατηγορίε. Τη 20 Οκτωβρίου του 2018 ο πρόεδρο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε την πρόθεση, είχαν την πρόθεση οι Ηνωμένε πολιτείε να αποσυρθούν από τη συνθήκη INF. Στις 26 Νοεμβρίου παραδέχθηκε η Ρωσία ότι είχε, ένα, είχε αναπτύξει ένα πύραυλο μέσου βεληνικού, ε, πύραυλο κρούζ το 9M729, αλλά επέμενε ότι ήταν κάτω από 480 χιλιόμετρα το βελινεκές, Επομένω ότι ήταν ε, σύμφωνο με τι διατάξεις της συνθήκης INF. 4 Δεκεμβρίου οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ εξέδωσαν μία διακήρυξη στην οποία κατέληγαν ότι η Ρωσία είχε αναπτύξει ένα πυραυλικό σύστημα και υποστήριζαν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, είχε δίκιο όταν έλεγε ότι παραβιάζει η Ρωσία τις υποχρεώσεις της βάσει της συνθήκης INF. Στις 2 Αυγούστου του 2019, οι Ηνωμένε Πολιτείε απασύρθησαν από τη συνθήκη INF, ενώ η Ρωσική Ομοσπονδία ε, είχε ήδη σταματήσει να εφαρμόζει τη συνθήκη. Παρά το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πολλές φορές ζητήσει από την Ρωσική Ομοσπονδία και πιο πρόσφατα στη διακήρυξη της ΥΠΑ εκπροσώπου της 14ης Ιουλίου να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν επανειλημμένα για την ανάπτυξη δοκιμή εν πτήση και ε, εγκατάσταση των, ε, του πυραυλικού συστήματος 9M729 και τις σοβαρές ανησυχίες για την ε, μη συμμόρφωση με τη συνθήκη INF. Όσον αφορά τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ε, καθεστώς που θα ισχύσει για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων μετά τη συνθήκη INF, Θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από όλα τα κράτη να κρατήσουν την ακαιρεότητα του διεθνού συστήματος ε, και βασική αρχή να είναι η αποτελεσματική πολυμέρεια. Αυτό είναι απαραίτητο για να κρατήσουμε τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Μας ενισχύει ότι το διεθνές Καθεστώ αφοπλισμού και μη διάδοση ε, βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση. Και α έχουμε κατά νου το διεθνές πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον για την ασφάλεια και τονίζουμε την ανάγκη να κρατήσουμε όλες τις πτυχές του αφοπλισμού και της μη διάδοσης για να βελτιώσουμε την παγκόσμια ασφάλεια. Οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να τηρούνται και να επιβάλλονται. Επαναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την δέσμευσή της για επαληθεύσιμους και αποτελεσματικούς ελέγχους με βάση τη συνθήκη και ενθαρρύνουμε την διατήρηση των επιτευγμάτων της συνθήκης INF. Δεδομένης της υψηλής έντασης, πρέπει να προσέχουμε να μην μπούμε σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών που θα αντιστάθμιζε τις σημαντικές μειώσεις που επετέφθησαν μετά το τέλος του πολέμου. Ενθαρρύνουμε λοιπόν τις ΗΠΑ και τη Ρωσική Ομοσπονδία να προσπαθήσουν να μειώσουν ε, τα, τον οπλισμό τους και τα στρατηγικά και τα μη στρατηγικά όπλα, τα οποία ε, είτε έχουν αναπτυχθεί είτε δεν έχουν αναπτυχθεί, λαμβάνοντα υπόψη την ειδική ευθύνη που έχουν οι χώρες που έχουν τα μεγαλύτερα ε, οπλοστάσια. Θέλουμε να αρχίσει ενεργός διάλογος για το μέλλον της συνθήκης ε, New Start μετά το 2021 δηλαδή, καθώς και για άλλες ρυθμίσεις για τον έλεγχο των εξοπλισμών. Και είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η συνθήκη New Start αποτελεί συνεισφορά στην υλοποίηση των υποχρεώσεων για τον αφοπλισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 της συνθήκης NPT για την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένωση υποστηρίζει τη συνθήκη ε, NPT για τη μη διάδοση των πυρηνικών ως ακρογωνιαίο λίθο ε, του παγκόσμιου καθεστώτος για τη μη διάδοση των πυρηνικών που είναι σημαντικός θεμέλιος λίθος ε, για να επιτύχουμε πυρηνικό αφοπλισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 της NPT. Η NPT παραμένει βασικό εργαλείο πολυμερούς ελέγχου που συνεισφέρει στη διεθνή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα. Αποτελεί μια ιστορική επιτυχία και η πλήρη υλοποίησή της απαιτείται τώρα περισσότερο από, από ποτέ. Θέλουμε να βελτιώσουμε το γενικότερο στρατηγικό περιβάλλον για τον αφοπλισμό, τη μη διάδοση και τον έλεγχο των εξοπλισμών για να σταματήσει η διάβρωση του διεθνούς συστήματος. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ε, ζητούμε από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της NPT να αρχίσουν ένα ε, επικοδομητικό διάλογο με σημαντικές προσπάθειες ώστε η διάσκεψη για την αναθεώρηση της συνθήκης NPT το 2020 ε, να είναι μια επιτυχία που θα αποτελέσει και ορόσημο μετά τα 50 χρόνια της συνθήκης. Ζητάμε από όλες τις χώρες που δεν έχουν υπογράψει και επικυρώσει ακόμη τη συνθήκη CTBT για την απαγόρευση των πυρηνικών να υπογράψουν και να επικυρώσουν το συντομότερο δυνατόν. Όσο εκρεμεί η έναξη ισχύω τη συνθήκη CTBT, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από όλα τα συμβαλόμενα μέρη να διατηρήσουν το μορατόριο για, τα πυρηνικά, για τις δοκιμές πυρηνικών όπλων ή οποιασδήποτε άλλες ε, χρήσεις πυρηνικών και επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δέσμευσή της ε, υπέρ των επαληθεύσιμων ελέγχων πυρηνικού αφοπλισμού και ελέγχου των όπλων και τονίζουμε την ανάγκη να ενδυναμώσουμε τον πολυμερή διάλογο και διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα τη διάσκεψη για τον αφοπλισμό. Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι απαιτούνται άμεσες διαπραγματεύσεις για μια συνθήκη που θα απαγορεύει την παραγωγή σχάσιμων υλικών για πυρηνικά όπλα ή άλλα ε, συστήματα πυρηνικών όπλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Αλμπέρκ. Μετά και εν ώψη των καινούριων ε, πυράβλων που ανέπτυξε η Ρωσία μετά την λήξη της συνθήκης, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το ΝΑΤΟ, εσείς κύριε Αλμπέρκ, πώς βλέπετε το μέλλον της μη διάδοσης των πυρηνικών σε που δεν θα παραταθεί η ισχύ της ε, συνθήκης. New start. Πάντοτε, πάντοτε αισθάνομαι ευγνώμη που έρχομαι εδώ να σας ε, μιλήσω. Δεν ξέρω αν θα σας εκπλήξει το ότι οι θέσεις της ε, ε, Ένωσης είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τις θέσεις του ΝΑΤΟ για την μη διάδεστα, πυρηνικά κλπ. Συμφωνούμε πάρα πολύ. Όμως, για να δούμε τι γίνεται πρώτα-πρώτα με το INF και κατόπιν να δούμε πώς βλέπουμε το μέλλον για τα πυρηνικά και τη μη διάδοση. Υπήρχε πολύ συγκεκριμένος ε, στόχος για τους SS-20. Πρόκειται για πυραυλό που οδήγησε τον ε, Σμιτ, τον καγκελάριο της Γερμανίας, να πει για απειλή, να κάνει αγόρευση σχετικά με την απειλή και έτσι ο στόχος ήταν να μην ισχυροποιηθεί η Ευρώπη και να δούμε το ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν αποσύρει τους και έκαναν καλύτερους οι Σοβιετικοί οπότε ο Σμιτ το 1977 στην συνάντηση κορυφής στο Λονδίνο είπε ότι θα πρέπει να εξισορροπηθεί αυτή η σοβιετική ισχύ, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση σε επίπεδο εξοπλισμών. Και από τα ανατολικά ουράλια μπορούσαν να χτυπήσουν στόχους στην ε, Ευρώπη. Οπότε αυτό ήταν μια πραγματική κρίση για την ε, Ευρώπη. Οπότε ήταν πάρα πολύ στριμωγμένο το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι. και όλα αυτά ήταν ε, διαβαθμισμένες πληροφορίες τότε δεκαετία του 70 τότε που υπήρχε αυτή η προβληματική για το πώς θα αντιδρούσε η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε. οπότε θα πρέπει να δούμε ότι ε, δεν θα ήθελε οπωσδήποτε να κάνει πόλεμο η Σοβιτική Ένωση. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε να πετύχουμε τον έλεγχο των εξοπλισμών. Να δούμε πώς θα υπάρχει αποτροπή της Σοβιετικής Ένωσης και οπότε είχαμε μια ειδική ομάδα για να σκεφτεί τι, τι μπορεί να γίνει. Θα δούμε... Ε, έχουμε την απόφαση του 79 και τη δήλωση για την ανάπτυξη των πυράβλων. Είπαμε ότι υπήρχε συγκεκριμένο αίτημα για την κατάργηση ε, αυτών των πυράβλων. Και άρχισαν οι διαπραγματεύσεις, το πήγαινε έλα και όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Γκορμπατζόφ συνέχισε τις συνομιλίες που είχαν διακοπεί και στο Ρεκεβίκη και Νέντσης κορυφής που αποτέλεσε μια επιτυχία, μια διέξοδο το αδιέξοδο και ξέρετε τι έγινε μετά το Δεκέμβριο του 87 σε να ισχύει αυτή η συνθήκη. Το 1987 και η περίοδος καταστροφής, κάτσε μέχρι το 91, ε, δεκαετής προειδοποίηση, επιθεωρήσεις. Και το 2007 ο Πούτιν είπε ότι δεν συνέφερε η INF την Σοβιετική Ένωση και το 2000 ε, επίσης, rocket forces in, the, in Russia in 2000, uh, Commander Yakolev said in the open Russian press that INF was not in Russia's interest. Και επίσης και άλλοι αξιωματούχοι σοβιετικοί άρχισαν να κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι παραβιάζονται συνθήκη και το ίδιο και ο Υπουργός Ιβάνοφ. Το ίδιο έγινε και στη συνέχεια το 2007 από τον ε, Πούτιν και τον, ε, τον Υπουργό Ιβανόφ. Οπότε, αυτά τα συστήματα των πυράβλων τι ωφελούν ακριβώ όπως οι ΕΣΕΣ. Πρόκειται να διχάσουν τους σύμμαχους ε, την Ευρώπη από τις ΗΠΑ και ξέρετε ότι το ΝΑΤΟ πάντοτε συμπαρατάσσεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Δεκέμβριο, το Φεβρουάριο είπαμε ότι στηρίζουμε τις Αμερικανικές αποφάσεις, αυτό είναι δύσκολη απόφαση, δεν θέλαμε να λήξει η συνθήκη. Και βέβαια, όταν η μία πλευρά περιορίζεται και η άλλη όχι, τότε αυτή η συμφωνία δεν βοηθά την ασφάλεια, αλλά υπονομεύει και τον έλεγχο των εξοπλισμών. Τότε η εισαβολιά αμείβεται. Ε, κάνει τη ζαβολιά ένας και αμείβεται γι' αυτό αντί για τον άλλο. Οπότε τα καλά νέα είναι ότι πριν από τέσσερα χρόνια ε, έχουμε καλά και κακά τέλο πάντων. Οι σύμμαχοι ενδιαφέρονται να μην συνεχιστεί ε, ο εξοπλισμός με τα πυρηνικά, έχουμε μη διάδοση. Το είπαν αυτό, το είπε το είπαν και το υπεστήριξαν και άρχισε στην Βιέννη ο διάλογος ε, στον φορέα για συνεργασία στην Ευρώπη και θέλαμε να υπάρχει διαφάνεια και όμως για κάποιο διάστημα ενώ υπήρχε ο διάλογος δεν έγινε τίποτα ουσιαστικό και συνεχίζεται ο διάλογος το 2014 επίσης. Συνεχίστηκαν κάθε χρόνο οι συναντήσεις και τον Δεκέμβριο πέρσι ήρθε ο υπουργό Ρώσος να μιλήσουμε τι γίνεται για όλα αυτά, για το Αφγανιστάν, για την Ουκρανία. Ε, είπα και Ρωσία στην Πράγα, στην Γενέβη, συνέχισαν τις επαφές και συνεχίζεται ο διάλογος για το καινούριο start και έχουμε και την διμερή επαφή, σύγχρονη την διμερή επι, επιτροπή. Συνεχίζεται επομένω ο διάλογος και έτσι συνεχίζονται η, η απειλή και η πίεση όσον αφορά το καθεστώς της μη διάδοσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και τώρα θέλουμε να δούμε τι θα γίνει στο επόμενο συμβούλιο με τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να θέλουν τον διερωτρομενό διάλογο. Την περασμένη εβδομάδα στον, ε, στη Βιέννη δουλέψαμε γι' αυτό. Έγιναν κάποιες επαφές και συζητήσαμε. Επόμενος γύρος ε, σύντομα θα γίνει και ό,τι και να σας πω είναι λίγο για το πόσο σημαντικό θεωρούμε το θέμα. Πρόκειται για την 50η επέτειο της ε, συνθήκης αυτής. Το 70 τέθηκε σε ισχύ. Η παράταση της συμφωνίας ήταν ε, κάτι που συνέβαλε στην ασφάλεια. Αποτρέψαμε 25 κράτη να αποκτήσουν πυρηνικά. Επομένω είναι βασική συνθήκη για αφοπλισμό και για ειρήνη παγκόσμια. Αυτό κάνει η συμμαχία. Και θέλουμε να πετύχουμε τους ε, στόχους μας αυτούς. Συνεχίζουμε να βοηθούμε ε, κάθε προσπάθεια προς ε, περισσότερη ασφάλεια. Ήταν ε, αρκετό στο παρελθόν να περιορίζεται η Ρωσία και είπα τώρα όμως έχουμε 20 χώρες που έχουν ε, πυράβλους. Προχωρημένη τεχνολογία και άρα πρόκειται για παγκοσμία απειλή. Θα πρέπει όλοι μαζί κάτι να κάνουμε. Θα πρέπει να θωρακίσουμε αυτά που έχουμε συμφωνήσει, αυτό το καθεστώς δεν θα πρέπει μόνο, είπα, και η Ρωσία να προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση, όλοι όσοι έχουν τις σχετικές τεχνολογίες. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται και με τα συμβατικά όπλα. Συμφώνησε η Συμμαχία, ούτως ώστε το έγγραφο της Βιέννης να αναθεωρηθεί εκ βάθρων. Sorry. That's my time being up. Α, χτύψε το ξυπνητήρι, έληξε ο χρόνος μου. Περιμένω τις ερωτήσεις σας. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Bruno pour... Euh, και τώρα το λόγο θα έχει ο κύριος Λετέ που θα μας πει για το τι επιλογές υπάρχουν στα όσα ισχύουν σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο και σας συγχαίρω και εγώ για την εκλογή σας ε, ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Εμείς ευχαριστώ, θα συνεργαζόμαστε μαζί σας. Δεν θέλω να μπω σε πολλά ιστορικά στοιχεία, αλλά ξεκινώντα την παρέμβασή μου, θέλω να σας υπενθυμίσω γιατί η συνθήκη INF αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ασφάλεια. Ήταν η συνθήκη που σταμάτησε την κρίση των πυράβλων μεταξύ ΙΠΑ και Ρωσία από το 1975 μέχρι το 1985. Και αυτή η κρίση κλιμακώθηκε τόσο πολύ που όταν υπεγράφει το 1987 η συνθήκη INF περίπου 3.500 πύραυλοι μέσω βεληνικούς τον είπα και της Ρωσίας απενεργοποιήθηκαν και αυτοί οι πύραυλοι ήταν πύραυλοι που ήταν στραμμένοι προς την Ευρώπη. Ξεκίνησα με αυτή την υπενθύμηση για να σας υπενθυμίσω περί τίνος συζητάμε δεν συμφωνούν η ε, Ρωσία και η ΕΠΑ σχετικά με τους πυράβλους και το ότι δεν συμφωνούν για την Ευρώπη αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ανησυχίες των τελευταίων 25-30 χρόνων. Εάν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν εκ νέου τέτοιους πυράβλους, η Ευρώπη βρίσκεται στη γραμμή του πυρός. Γι' αυτό οι στρατηγικές συζητήσεις είναι πολύ σημαντικές είτε μπορούμε να ξεφορτωθούμε αυτά τα όπλα, είτε θα στραφούν και πάλι ε, στοχεύοντας προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είναι μια πολιτική επιλογή λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να οθεί και του Αμερικανού και του Ρώσους να συνεχίσουν τι προσπάθειε προ τον έλεγχο των εξοπλισμών ή ακόμη καλύτερα προ τον αφοπλισμό. Διότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον να κινηθούν προ τέτοιε συζητήσει. Εμεί, λοιπόν εδώ στην Ευρώπη πρέπει να ενθαρρύνουμε τι δύο πρωτεύουσε να ξεκινήσουν τέτοιε συζητήσει. Και για να πούμε την αλήθεια δεν θα είναι καθόλου εύκολο αυτό. Με το τέλος της συνθήκη INF δεν υπάρχει ένα εναλλακτικό σενάριο σε ολόκληρο τον κόσμο για τον έλεγχο των πυράβλων μέσου βεληνικούς, ούτε υπάρχει και κάποια προοπτική για ένα δεύτερο σενάριο στο προσεχές μέλλον. Είμαι λοιπόν διστακτικός ε, για το τι μπορεί να γίνει. Ο έλεγχο των εξοπλισμών, και εδώ ίσω να διαφωνώ λίγο με τον ε, συνομιλητή που έλεγε το λόγο πιο πριν, ε, δεν δεν είναι πια παλιωμοδίτικη η συνθήκη και πρέπει να σκεφτούμε τι είδους συνθήκες μπορούμε να έχουμε σαν τη νέα συνθήκη START. Και ο Αντώνιο Γκουτιέρες, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, είπε ότι ο κόσμος ε, έχασε αυτό το πολύτιμο διάλειμμα το οποίο είχαμε ε, μετά τον ψυχρό πόλεμο. οι στρατηγικές ανησυχίες που έχουμε πρέπει να συζητηθούν για να καταλάβουμε και τις διάφορες παραμέτρους για το μέλλον. Όσον αφορά ε, τη Ρωσία, δεν υπάρχει καμία στρατηγική αξία, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τη διατήρηση της συνθήκης INF. Η Μόσχα δαπανά σημαντικά κονδύλια για την ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων Cruise. Έχει ήδη αναπτύξει δύο SSC8, μία στο Εκατερίνεμπουργκ και μία κοντά στο κάπου στην Τζάρ, στην Κασπία. Η χρήση πυράβλων μέσου βελνικούς είναι κομμάτι της ε, στρατιωτικής τακτικής της Ρωσίας. Είναι τα ενεργά μέτρα που συνδυάζουν υβριδικά ε, όπλα και πυρηνικές δυνάμεις για να αποσταθεροποιήσουν τους αντιπάλους. Επομένως, ε, η συνθήκη INF είναι αντίθετη με τις στρατηγικές επιδιώξεις της Ρωσίας. Δεύτερον, αν δούμε την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραμένουν υπέρμαχοι του ελέγχου των εξοπλισμών, προσπάθησαν να υπερασπίσουν τη συνθήκη INF όσο μπορούσαν, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι η συνθήκη άρχισε να γίνεται οριακή για τα συμφέροντα των Αμερικανών. Και γιατί? Καταρχήν, διότι υπάρχει ένα σαφές ε, σημάδι ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να επενδύσει σε πυράβλους μέσου βεληνικούς για να υπερασπίσει τους ε, συμμάχους της ε, στην Ασία από απειλές σε αυτή την περιφέρεια και υπάρχει ε, η πρόθεση να εγκατασταθούν πυρηνικές κεφαλές σε υποβρύχια που κινούνται στην περιοχή ε, ε, εκείνη. Αυτό δεν ήταν εύκολο να γίνει με τη συνθήκη INF. Δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αντίστοιχοι πύραυλοι στην Ευρώπη και τώρα χωρίς την συνθήκη INF μπορούν να εγκατασταθούν ε, μπορούν ε, να συνεχίσουν να υπάρχουν στη Ρουμανία οι εκτοξευτές και τα συστήματα αυτά που είναι αμυντικά μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε επιθετικά. Το Φεβρουάριο του 2018 στην αναθεώρηση της πολιτικής τους αναφέρεται σαφώς αυτή η προοπτική. Ε, τρίτον, και η Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να απελευθερωθούν από τις δεσμεύσεις της συνθήκης, γιατί έχουν διαπιστώσει ότι νέες απειλές υπάρχουν στην Νοτιοανατολική Ασία, Νότια, Βόρεια Κορέα, Πακιστάν, Κίνα και οι απειλές αυτές αυξάνονται εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Η Κίνα έχει αναπτύξει το πλωστάτιό τη με πυράβλου μέσου βελληνικού, γιατί ποτέ δεν ήταν συμβαλόμενο μέρο, μέρος της συνθήκη INF. Και η Μόσχα και η Ουάσιγκτον αυτό το θεωρούν στρατηγικό μειονέκτημα. Η απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αποχωρήσει από τη συνθήκη INF ε, ε, ελήφθη στο πλαίσιο των γενικότερων, ε, της γενικότερης κατάστασης που περιλαμβάνει και την Κίνα. Βέβαια οι Κινέζοι αντέδρασαν έντονα, είπαν ότι δεν θα πρέπει οι Ηνωμένε Πολιτείε να εκβιάζουν την Κίνα. Αλλά το 90% των εκτιμόμενων 1.600 πυράβλων κρούς της Κίνας είναι μέσα στο βεληνικές της συνθήκης INF. Αν λοιπόν είχε υπογράψει μια τριμερή συνθήκη INF η Κίνα, θα είχε χάσει όλο της το δυναμικό που την κάνει ισχυρή δύναμη στην περιφέρεια του μέσου ελληνικού. Άρα δεν νομίζω ότι είναι πιθανό να μπει σε μια τέτοια συμφωνία η Κίνα. Για να δώσω τώρα μια γενικότερη επισκόπηση αυτών των στρατηγικών ε, ε, επισκοπήσεων, ε, θέλω να πω ότι η συνθήκη INF ίσως ήταν παροχημένη τα τελευταία χρόνια. Οι Ηνωμένε Πολιτείε άρχισαν σχέδια για δοκιμές ενός νέου μη πυρηνικού συμβατικού πυράβλου Cruise, προκαλώντας ε, ε, συγκεκριμένα τη Ρωσία και την Ευρώπη. Το Πεντάγωνο είπε ότι τέτοιοι καινούργοι πύραυλοι μπορούν να είναι έτοιμοι να αναπτυχθούν μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Αρχές του 2021 δηλαδή θα μπορούσαν να είναι έτοιμοι. Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε 96 εκατομμύρια δολάρια το 2020 ως προϋπολογισμό για να συνεχίσει την έρευνα για πυράβλους που καλύπτονται από το βεληνικές της πρώην συνθήκης ε, INF αν προχωρήσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε στην ανάπτυξη βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων κρούζ, το βασικό ερώτημα παραμένει πού θα αναπτυχθούν αυτά τα συστήματα. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, Υπάρχει μια λογική στρατιωτική επιλογή ότι τέτοια συστήματα θα μπορούσαν ε, ταχαίως να αναπτυχθούν στην Ευρώπη. Διαφορετικά τέτοιοι πύραυλοι μέσου βελληνικούς δεν θα είχαν ε, δυνατότητα αποτροπής έναντι της Ρωσίας. Και εδώ ε, μπαίνει και ο ρόλος του ΝΑΤΟ. Πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε ένα θεωρητικό αίτημα των ΗΠΑ να αναπτύξει πυράβλους στην Ευρώπη. Σήμερα κανένα μέλος του ΝΑΤΟ δεν έχει πει ότι θα είναι πρόθυμο να έχει στο έδαφος του τέτοιους πυράβλους μέσου βεληνικούς. Αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ Μάλιστα, έχουν πει δημοσίω ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη τέτοιων πυράβλων στην Ευρώπη θα πρέπει να έχει εγκριθεί από όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Και ο Γενικό Γραμματέα Γιάννη Στόλτεμπεργκ είπε ότι θα πρέπει να γίνει ο συντονισμό μέσα στην οικογένεια του ΝΑΤΟ για τέτοια θέματα και όχι με διμερεί συμφωνίε. Υπό το φως όλων αυτών, λοιπόν, νομίζω ότι τρία σενάρια διαμορφώνονται για την Ευρώπη μετά την συνθήκη INF. Το πρώτο σενάριο είναι ότι μια Ενωμένη Ευρώπη ε, απορρίπτει την ανάπτυξη αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων στο έδαφος της, ε, αλλά αυτό θα διαβρώσει τις ε, διατλαντικές σχέσεις και δεν θα εμποδίσει τη Ρωσία να αναπτύξει τα δικά της συστήματα. Ένα δεύτερο σενάριο είναι ότι μια Ενωμένη Ευρώπη μπορεί να επιλέξει μια κούρσα εξοπλισμών ε, έναντι της Ρωσίας με υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι σαν ε, αυτό που συνέβη το 1975, με κάποιες διαμαρτυρίες από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Και ένα τρίτο σενάριο είναι ότι μπορεί να υπάρξει ένα σπισμός πρόθυμων ευρωπαϊκών χωρών που θα δεχθούν ανάπτυξη αμερικανικών πυράβλων στο έδαφος τους. Και αυτό θα διακινδυνεύσει να έχουμε ε, μια διάσπαση στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Καμία λοιπόν από τις τρεις λύσεις, ε, κανένα από τα τρία σενάρια δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για την Ευρώπη, αλλά είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας την τύχη μας. Οι επιλογές μας θα έχουν επιπτώσεις για την ασφάλεια των επόμενων γενιών, τουλάχιστον της επόμενης γενιάς. Επομένως, η Ευρώπη θα πρέπει να ασχοληθεί πολύ δραστήρια με αυτό το θέμα, γιατί αν δεν το κάνουμε, το τίμημα θα είναι ότι θα χάσουμε επιρροή σε ένα θέμα που έχει βασική σημασία για την ασφαλειά μας. Και θα πρέπει να δούμε τι κάνουν και άλλες μεγάλες δυνάμεις. Μήπως δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ήπειρος γίνει και πάλι ένα πεδίο μάχης ή ένα διπλωματικό ατού στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και απεσιόδοξη παρουσίαση και θα συνεχίσουμε δίνοντας τώρα το λόγο στους συντονιστέ που μου ζητήσει το λόγο. Πρώτα-πρώτα για το έλκο κύριο Ντονζό. Σα ευχαριστούμε κύριε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το να δούμε το ιστορικό πλαίσιο και το γεωγραφικό μας κυριολετέ και πρόκειται για μια καινούργια γεωστρατηγική και έτσι έχει αναδεθεί τώρα το σκηνικό ε, της Ασίας και πιο συγκεκριμένα της ε, Κίνας που αλλάζουν τα πράγματα σε σχέση με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού γιατί όπως μας ε, τονίσατε αυτό το ανησυχητικό θέμα όσον αφορά το πόσο κόντρα τη συνθήκη η Ρωσία αλλά και επίσης το καινούριο ζήτημα της αμερικανικής ανησυχίας σε σχέση με το τι γίνεται στην Ασία. Καινούργια αυτά στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη γιατί έχουν επίσης και τεχνική, τεχνοκρατική σημασία γιατί ίσως το ΝΑΤΟ δεν είναι ο σωστός τόπος ούτως ώστε να συζητάει η Δύση αυτά τα ζητήματα. Μιλάμε τι γίνεται στον Ειρηνικό, οπότε πια το ΝΑΤΟ εκεί δεν έχει αρμοδιότητα. Όσον αφορά όλα αυτά, την προβληματική της Δύση. Οπότε ε, αποκομίσαμε ως εντύπωση από είπατε ότι κανείς από τους βασικούς παράγοντες η ε, Κίνα, Ρωσία δεν έχει συμφέρον ούτω ώστε να αναδεθεί ξανά η συνθήκη με την μορφή που είχε ε, εμείς όμως οι Ευρωπαίοι και για αυτό το θέμα όπως και για άλλα δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε γαντζωμένοι ακόμα στο παρελθόν όσον αφορά την πολυμερή μέθοδο. Ε, εντάξει, υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι γιατί έχουμε αυτό την κατάρρευση όλων αυτών των δομών, δεν μπορούμε αυτό να το παρακάμψουμε, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχουμε καταλήξει σε κάποια plan B, ούτως ώστε να υπάρχει μια άλλη αρχιτεκτονική. Και ακριβώς εδώ νομίζω ότι πάσχει η δική μας θέση. Θα πρέπει να εξωθήσουμε τους ε, διεθνείς παράγοντες να τα βρούνε, να βρούνε τα μέσα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι κανένας από αυτούς τους διεθνείς παράγοντες δεν το θέλει. Οπότε εμείς δημιουργούμε την εντύπωση αυτή ότι είμαστε κολλημένοι σε κάτι που είναι πια ξεπερασμένο. Παρατήρησα αυτό, δεν είναι ερώτηση, αλλά τέλος πάντων είναι τα πράγματα σκούρα, αυτό διαπιστώνουμε σε σχέση με αυτά τα σενάρια που μας ε, εξήγησε ο κύριος Λετέ και ελπίζω ότι όλα αυτά δεν θα υλοποιηθούν που μας είπατε αλλά σήμερα συνειδητοποιώ ότι σε σχέση με την ανάπτυξη την ενδεχόμενη των Αμερικανικών πυράβλων έχουμε τις διμερείς συνθήκες γιατί βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη τι γίνεται σε σχέση με το απρόβλεπτο της Αμερικανικής κυβέρνησης, του Προέδρου συγκεκριμένα ότι έχουμε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών που πηγαίνουν μόνες τους να μιλήσουν στην Ευρώπη, στην Αμερική, συγγνώμη, στην Ουάσιγκτον, διμερός. Ε, αυτό <clears throat> είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί αυτό δίνει την ε, πρόφαση στους Ρώσους. Να πούνε, να, δεν έχει αξιοπιστία το ΝΑΤΟ. Οπότε, εγώ εκεί, εκεί μένω, σε αυτό το απεσιόδοξο σενάριο που μας εξηγήσατε. Μπράβο όμως για την ε, παρουσίαση της παρουσιάσεις σας που ήταν τόσο πλήρες και μας εξηγήσατε το πόσο στριμωγμένοι έχουμε βρεθεί σήμερα. Και να δούμε τι, πώς, πόσο θετικά είναι τα σενάρια, τα πρόθεσμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσιάση σας. Είναι δύσκολο το δίλημα αυτό στο οποίο βρισκόμαστε όταν μιλούμε για την ευρωπαϊκή προσέγγιση του, απέναντι στο θάνατο της INF. Ε, ίσως να προτιμούμε τις ε, πολυμερείς ε, δραστηριότητες καλύτερα από τις διμερείς και τις συμφωνίες και σίγουρα δεν θα θέλαμε να καταργηθεί μια υπάρχουσα διεθνή διμερή συμφωνία επειδή μόνο και μόνο δεν υπάρχει κάτι να την αντικαταστήσει στο εγγύς μέλλον ή στο άμεσο μέλλον. Αλλά Δεχόμαστε και το επιχείρημα τον είπα ότι δεν έχει και πολύ νόημα να πρέπει κανείς να παραμένει σταθερό στα δικά του, στις δικές του απαιτήσει αν το άλλο μέρος της διμερούς συμφωνίας παραβιάζει αυτούς ακριβώς τους όρους της συμφωνίας. Υπάρχουν τρία σενάρια τα οποία μας διαβάσατε. Τα δύο μάλλον δύσκολα θα επιτευχθούν. Η ομοφωνία στο ΝΑΤΟ η συγκατάθεση για την αποδοχή της Αμερικανικής Ανάπτυξης ή της απόρριψης του αιτήματο των ΗΠΑ μάλλον δεν θα περάσει πολύ εύκολα σε σχέση με την ε, ε, με τις διμερείς συμφωνίες. Και ίσως αυτό δεν ε, είναι και πολύ διαφορετικό μετά από τα όσα έγιναν ε, όταν εξέπνευσε η συμφωνία ABM, όταν αρχίσαν οι διάφορες χώρες να διαπραγματεύονται τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για τα διάφορα αντίστοιχα συστήματα των πυράβλων και τα αμυντικά. Και το ερώτημά μου είναι, κυρία Αλμπέρκ, αναφέρατε διάφορα συστήματα ε, ελέγχου των όπλων και, συμφωνιών, και συμφωνίες που ε, βρίσκονται ε, εν κενό. Τα όσα έχουν γίνει στη Βουδαπέστη δεν έχουν ολοκληρωθεί όμως, μετα, δηλαδή εκ των πραγμάτων μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας. Και επίσης αυτή η νέα συμφωνία New Start. Είναι ενθαρρυντικό που συνεχίζονται οι συζητήσεις μετά την συμφωνία αυτή. Αλλά τι θα γίνει ακριβώς εάν δεν ολοκληρωθούν αυτές οι συζητήσεις μέχρι να εκπνεύσει το 2021 όπως περιμένουμε η συνθήκη New Start. Θα εκπνεύσει αυτόματα το 2021 ή θα υπάρξει μια κατάσταση παραμονής της μέχρι να υπάρξει κάτι καινούριο. Και μετά θυμούμε ότι μετά την, ε, τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου εναντίον των ΗΠΑ το σενάριο των, του, του πυρηνικού υλικού που θα μπορούσε ίσως να πέσει σε λάθος ε, χέρια ήταν ένα ε, θέμα που το συζητούσαμε πολύ. Ε, έχει υποχωρήσει λίγο αυτή η ανησυχία, αλλά πάντα υπήρχε αυτή, πάντα, αλλά υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία για την ασφάλεια του πυρηνικού υλικού ή υλικού χάσει ή το, για την εξασφάλιση του ουρανίου, για να μην χρησιμοποιηθεί δηλαδή από λάθο χέρια για στρατιωτικού ή τρομοκρατικούς σκοπούς. Ε, εδώ τι γίνεται ακριβώς. Ευχαριστώ. Προτείνω στους τρεις ομιλητές να λάβουν το λόγο μετά από αυτές τις πρώτες παρατηρήσεις. δεν ήταν μόνο ερωτήσεις, ήταν παρατηρήσεις αρκετές. και είμαι βέβαιη ότι θα ξεκινήσουμε και με άλλες ερωτήσεις μετά από αυτά που έχετε να μας πείτε. Yes, thank you very much uh, for, for, for... Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και τις παρατηρήσεις. Λοιπόν, για το κατά πόσο εμείς στην Ευρώπη υποστηρίζουμε ε, ένα παλιό σύστημα που έχει πια εκπνεύσει ή παρέλθει. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό για τις μικρές ή τις μεσαίου μεγέθους χώρες να εμπιστεύονται τις πολυμερείς συμφωνίες μέσα σε αυτή την νέα τάξη πραγμάτων. Είναι φυσικό οι μικρές χώρες να αισθάνονται λίγο πιο κοντά στον πολυμερισμό, στην πολυμέρεια και στα και σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Και επίσης, το σύστημα που ε, υποστηρίζουν μας έχει δώσει και δεκα, δεκαετίες ειρήνης και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν ε, ακόμα καλά επιχειρήματα να επιμείνουμε στη διατήρηση αυτών των πολύτιμων στοιχείων και για τη μη διάδοση, όπως η συνθήκη που αναφέραμε. Βεβαίω αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι απορρίπτουμε νέες προτάσεις, νέε πρωτοβουλίες. Αλλά το σημαντικό που πρέπει να έχουμε σίγουρα υπόψη είναι ότι το καλύτερο μπορεί να είναι ο του καλού. Νομίζω ότι έχουμε και εμείς τις δικές μας προτάσεις σε διάφορους τομείς για νέες ε, ε, συνθήκες ή συμφωνίες, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνει ε, για, ε, πετώντας ό,τι καλό έχει γίνει μέχρι στιγμή. Πρέπει να βασιστούμε στα καλά και να συνεχίσουμε. Α πούμε, η, η νέα αυτή συνθήκη, New Start, θα σταματούσε να ισχύει αν δεν υπάρξει κάτι μετά από αυτή. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει κάτι πριν τη Δευτέρα Φεβρουαρίου του 2021, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει δηλαδή μέχρι τότε, τις 2 Φεβρουαρίου, να έχει υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων ε, μεταξύ Ουάσιγκτον και ε, Μόσχας για την παράταση για πέντε χρόνια. Έτσι, έχουμε το χρόνο να, διαπραγματευτούμε περαιτέρω. Σίγουρα οι διαπραγματεύσει στον τομέα αυτό παίρνουν χρόνια, είναι ούτως ή άλλως περίπλοκες. Μετά, το μνημόνιο της Βουδαπέστης, νομίζω θα το πει ο συνάδελφος, ε, τα, ε, τα σενάρια τώρα για τις βρώμικες βόμβες, ε, νομίζω ότι και οι δύο μας οργανώσεις επικεντρώνονται πολύ σε τέτοιου είδους σενάρια. Στην Ευρώπη, πρώτα κοιτούμε την ενίσχυση των νομικών συστημάτων βέβαια. Υποστηρίζουμε, ας πούμε, την ε, ε, αποτελεσματική εφαρμογή της τροποποιημένης συνθήκης για την φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού, την Διεθνή Σύμβαση για, τον πυρηνικό, για την πυρηνική τρομοκρατία. Ε, συνεργαζόμαστε με το Αγραφείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε μια καθολική εφαρμογή και να έχουν οι χώρε τι δυνατότητε να εφαρμόζουν τέτοιου είδου νομικέ συμφωνίε. Αλλά επίση κάνουμε και δουλειά επιτόπου όπως ας πούμε με τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας. Αυτή η πρωτοβουλία είναι παγκόσμια ε, πρωτοβουλία για τη δημιουργία δυνατοτήτων στις τρίτες χώρες, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε πολλά σενάρια χημικών, ε, βιολογικών, ε, ραδιενεργών υλικών κτλ. όχι μόνο δηλαδή ατυχημάτων και τρομοκρατικών επιθέσεων. Και επίσης συνεργαζόμαστε φυσικά και πολύ στενά με το ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Για το πρώτο σχόλιο, το εκτιμώ. Το ΝΑΤΟ όντω δεν είναι το βήμα για να λύσουμε τα προβλήματα των πυράβλων παγκοσμίων, αλλά οι σύμμαχοι μπορούν να συμβάλλουν και έχουμε συζητήσεις ε, με την Αυστραλία, την ε, Νότιο Κορέα, την Ιαπωνία, ακόμα και με την Κίνα κάνουμε συζητήσεις. Και εγώ προσπαθώ να οργανώσω άμεσα, ε, άμεσο κανάλι επικοινωνίας με την Κίνα, με το ΝΑΤΟ. Αλλά ο τελευταίος γύρος του κώδικα δοντολογίας για τις για τους πυράβλους ε, συμπληρώθηκε από τη Γερμανία που είχε πολύ καλές προτάσεις. Και πρέπει βεβαίω να ξέρουμε ποιο θα πάει σε αυτή, την, ε, σε αυτή τη συνάντηση για να ξέρουμε πώ θα, την, ε, πώς θα προετοιμαστούμε. Πρέπει, ας πούμε, να μοιραστούμε οι σύμμαχοι της απόψει μα και μετά να πάμε με 40-50 χώρε και να πούμε εδώ είμαστε, θέλουμε να ενισχύσουμε τους ελέγχους των πυράβλων. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε λίγο περισσότερο ζήλο λίγο περισσότερες προτάσεις στο Καθεστώ ε, ελέγχου, ε, το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια, υπάρχει ο, ο δοντολογία δοντολογίας επιτάπητος, αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση χωρών. Όπως είδαμε και για την ε, PCW. Όταν οι χώρες πιέζουν και θέλουν να πιέσουν στο ανώτατο επίπεδο, επιτυγχάνονται αποτελέσματα. Και βεβαίως πρέπει να υπάρξει και μια νέα, ένα νέο παγκόσμιο σκεπτικό η ε, Κίνα σίγουρα δεν θα ε, συμφωνήσει να καταργηθούν όλοι οι πύραυλοι, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε, ε, ας πούμε, για του μη βαλιστικού πυράβλους κάποια διαφάνεια. Νομίζω ότι μπορούμε να πιέσουμε. Η νέα αυτή συμμαχία, λοιπόν, και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για τέτοιου είδου δημιουργία μια παγκόσμια συμμαχία να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδου απειλέ. Εγώ τουλάχιστον ω προ αυτό δουλεύω. Και σε σχέση με τα εξαιρετικά σχόλια που κάνατε εσείς, Πρέπει να θυμόμαστε ότι τότε η συνθήκη INF ήταν ένα βήμα σε μια αλληλουχία βημάτων. Η συμμαχία του ΝΑΤΟ κάλεσε τη Σοβιετική Ένωση να μετατρέψει τις ε, ε, ε συζητήσεις ε, και να ξεκινήσει συζητήσεις για τους πυράβλους ε, αυτό ήταν δηλαδή το επόμενο βήμα. Αλλά επειδή κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, δεν φτάσαμε ποτέ σε αυτό το στο επόμενο βήμα. Όταν, η συνθήκη, όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει τη συνθήκη INF, οι ΗΠΑ είχαν ε, ε, πάρα πολλού κρούζ ε, πυράβλου και όταν τελείωσαν οι διαπραγματεύσει είχαν αντίστοιχου και οι Ρώσοι. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε τώρα, αυτό που ήταν το σκεπτικό των ε, υπερδυνάμεων, τώρα είναι το σκεπτικό μεγάλων εταιριών. Οπότε πρέπει να παγκοσμιοποιήσουμε και εμεί λίγο το σκεπτικό μα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αν, αν συμφωνήσουν οι ΗΠΑ με τη Ρωσία για την συνθήκη θα λυθούν τα προβλήματα όλων. Πρέπει να τα δούμε τα θέματα αυτά σε πιο ευρύ πλαίσιο. Και για το μνημόνιο τη Βουδαπέστη η παραβίαση της ε, Ρωσίας είναι ξεκάθαρη του μνημονίου αυτού. Αυτό ήταν η υπόσχεση του Ηνωμένου Βασιλείου, ήπα Ρωσίας και Γαλλίας στην Ουκρανία, στην Λευκορωσία και στο Καζακστάν να καταργήσουν τα πυρηνικά όπλα και να μπουν στη σύμβαση ω μη πυρηνικέ χώρε. Με αντάλλαγμα μη οικονομική πίεση, πολιτική πίεση ή αλλαγή συνόρων. Η Ρωσία τα καταπάτησε όλα αυτά. Αλλά αυτέ οι υποσχέσει εξακολουθούν να υπάρχουν. Η Ρωσία βεβαίω μπορεί να τι ξανακαταπατήσει, μάλιστα τι καταπατά τώρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ε, έχουν καταπατηθεί από τι υπόλοιπε χώρε αυτέ οι συμφωνίε, οι υποσχέσει. Εξακολουθούν να είναι και μέλο των ε, δικλειδών ασφαλεία του ΝΑΤΟ. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι οι εγγυήσει των άλλων χωρών εξακολουθούν να είναι ε, ενισχύει. Και θα πρέπει φυσικά. Τώρα, για το υλικό το πυρηνικό. Μιλήσατε για κάποιε από τις ε, εξελίξεις για, τον ε, για την πυρηνική τρομοκρατία. Υπάρχουν ε, οι διάφορες σύνοδοι κορυφής που, που έκανε και ο πρόεδρος Ομπάμα. Υπάρχει το ψήφισμα 1540. Οπότε μπορεί να μην, έχει, να μην το βλέπουμε σε πηχαίους τίτλους της ειδήσει, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πράγματα που γίνονται ώστε να φύγουν τα, υλικά αυτά από επικίνδυνους και το θέμα είναι να μην υπάρχει ε, πρόσβαση από μη ε, κρατικούς φορεί σε χημικά για να τα χρησιμοποιήσουν. Α πούμε στη Συρία ή στην ε, Βόρεια Κορέα τα χημικά όπλα είναι πάρα πολύ σημαντική ανησυχία. Και όσοι δεν είναι κρατικοί φορεί, βλέπουμε να αποκτούν ξαφνικά όπλα μη πυραυλικά και δυνατότητε. Αντίστοιχε. Αυτά από μένα και σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να απαντήσω ε, καταρχήν σε αυτά που είπε ο κ. Ντανζό γιατί λίγο πολύ συμφωνώ μαζί σας για τη συνθήκη INF, παραδείγματο χάρη. Και εγώ νομίζω ότι εμείς στην Ευρώπη θέλαμε να τη σώσουμε, αλλά δεν θέλανε πολύ σε όλο τον κόσμο να σωθεί η συνθήκη INF τελικά. Μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής μας για την ασφάλεια στην Ευρώπη βασίζεται σε συνθήκη, συνθήκες της δεκαετίας του 90. Ε, η συνθήκη INF, CFE, το Memorandum της Βουδαπέστης. Χρειαζόμαστε κάτι που να αντιστοιχεί στις πραγματικότητες τη σημερινές. Και οι πραγματικότητες είναι ότι έχουμε διαφορετικές συνθήκες και στι ΗΠΑ. η Ρωσία έχει ανακάμψει και βεβαίως ε, η Κίνα αναδύεται ως δύναμη. Αυτά που είχαμε λοιπόν ως συνθήκες στη δεκαετία του 90 πρέπει να τα εξυγχρονίσουμε πλέον και πρέπει να είμαστε πρακτικοί με ευέλικτες λύσεις σύμφωνες με την ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε. Επανέρχομαι τώρα στο θέμα μας που είναι το τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Αν ε, είχα τη δυνατότητα να προτείνω πολιτικές, γιατί εγώ είμαι μόνο ε, μεταξύ αυτών που θεωρητικά εξετάζουν το θέμα, ως πολιτική θα πρότεινα καταρχήν τη νέα συνθήκη START, που λύγει το 2021, δεύτερον πίεση στη Ρωσία σχετικά με τους πυράβλους μέσου ελληνικού και μάλιστα διτή πίεση με αποτροπή ασκήσεις κλπ που έχει ήδη προτείνει το ΝΑΤΟ κάτι τέτοιο, όπως επίσης και συνομιλίες με τη Ρωσία. Βέβαια το χρειαζόμαστε, παρότι θα είναι δύσκολες. Και η τρίτη προτεραιότητα είναι να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε διάφορα σενάρια. Αν οι πρώτες δύο λύσεις αποτύχουν, να διαμορφώσουμε κάποια σενάρια για την Ευρώπη και να είμαστε προετοιμασμένοι για τα σενάρια αυτά. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να είμαστε έτοιμοι είτε για επιτυχία είτε αποτυχία αυτών των σενάριων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, για τις απαντήσεις σας και για τα σχόλιά σας. Θέλει κάποιος άλλο το λόγο. Έχετε παρατηρήσεις. Κύριε Σατόρη. Merci, Madame la Présidente. Merci. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε για τις εισηγήσεις σας που ήταν ξεκάθαρες, βέβαια, όπως είπε ο Πρόεδρος, ανησυχητικές. Και σήμερα γινόμαστε μάρτυρες από αυτή την ε, πλήρη περιγραφή της κατάστασης της κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λύση, βέβαια μας υποδείξατε κάποιες λύσεις ε, στην τελευταία ομιλία. Αλλά αυτό θέλω να σας πω και να πω σε όλους τους αδελφούς εδώ και στην Πρόεδρο. Εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς μπορούμε έτσι να εκπονήσουμε μια στρατηγική της Ένωσης για αυτή την κατάσταση και τι πρωτοβουλίες που υπάρχουν τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, όλοι μαζί ως ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Ε, βέβαια, είναι φυσιολογικό να ανησυχούμε γιατί είμαστε αυτοί που περισσότερο ωφελούμε από τη, τα, τα, τα καλά, την προστασία της συνθήκης INF. Ναι, πολλές φορές Ε, βέβαια και είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής πολυμερούς ε, προσέγγισης ε, σε, σε κάθε επίπεδο, σε κάθε στρατηγική, εμπορική, οικονομική και στρατηγικά βλέπουμε. Αλλά διαπιστώνουμε ότι ε, υπάρχει τέτοια προσέγγιση και για τα θέματα του πυρηνικού αφοπλισμού. Το θέμα επίγει είναι η ασφάλεια των Ευρωπαίων και το ότι υπάρχει διάδοση των πυρηνικών και η πραγματική δυσκολία εκεί έγκυται ισχύει σήμερα η συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών, την εκπόνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, την πρόσυπέγραψαν, την εκείρωσαν μια σειρά κρατών μελών. Πώς, πώς και εμεί εδώ μπορούμε να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί στον κόσμο για το θέμα του πυρηνικού αφοπλισμού. Euh, δεν θέλει άλλο το λόγο, λέει η πρόεδρο, να απαντήσω εγώ. Μια που και σε μένα και σε... Καλά σε όλους μας απευθύνεται η ερώτηση. Ακούσαμε τις ε, εισηγήσει πολύ χρήσιμες. Ε, γιατί έτσι ε, καταλάβαμε τι κατάσταση έχουμε ενώπιόν μας, ιδιαίτερα ανησυχητική, κυρίως για την Ευρώπη και το πράγμα επιδέχεται και επιδίνωσε εάν δεν γίνει δίπλα με την συνθήκη Στάρτ. Ακούσαμε τι είπε ο Μπρίνο Λετέ, μας ε, υπέδειξε κάποιες λύσεις. για το τι στάση πρέπει να τηρήσουμε αντί της Ρωσίας. αποτροπή και διάλογος. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει την πολυεμερή μέθοδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε νοσταλγοί των συνθήκων που συνήφθησαν ε, σε άλλη εποχή, μια άλλη συγκυρία. Ιδίω για το ΑΙΑΝΕ θα πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχουν και άλλες συνθήκες αλλά το να θέλουμε την πολυμερή μέθοδο δεν σημαίνει ότι θέλουμε τον, την, την αδράνεια. Κίνα, Ρωσία είναι οι παράγοντες διεθνείς ε, σήμερα η ΕΠΑ και δεν είναι αυτή υπέρ της πολυμερίας. Τι πρέπει να γίνει. Εγώ ενδεικτικά θα ήθελα να πω ότι στην ακρόαση του Ζωζέ Μπορέλ κάποιος από μας να θέσει το ερώτημα. Τι προτίθεται να κάνει εάν καταρρεύσει η INF. Επίσης, οι συντονιστές να το συζητήσουν και σε μια συνεδρίαση να προγραμματίσουν τη δουλειά μας για το μέλλον. Για το θέμα αυτό του ελέγχου των εξοπλισμών, για το παγκοσμίο σύστημα του, του ελέγχου των εξοπλισμών, για τις συνθήκες να συνεχίσουμε τη δουλειά μας με τη βοήθεια των ειδικών και έτσι να επεξεργαστούμε κάποιες προτάσεις. Αυτά για τους συντονιστές. Αλλά δεν με εκπλήσουν αυτά τα οποία ακούσαμε που θα αποτελέσουν αφετηρία για τη δουλειά μας κατά αυτή την θητεία. Ευχαριστούμε και τους τρεις ομιλητές μας. Ήσασταν ε, σαφείς, ήσασταν ξεκάθαροι, ειλικρινείς. Έχετε το λόγο, κύριε Μπιαλίτσεκ. Ευχαριστώ. Τέτοιου είδου συζητήσει είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται και για εμά στην Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, για να έχουμε μία αίσθηση του ε, ποια είναι η κατεύθυνση και ποιο είναι το ενδιαφέρον που δείχνει το ε, Κοινοβούλιο και, στο και προς την οποία θέλει να δουλέψουμε. Έχουμε και την σχετική ομάδα εργασία, ε, η οποία ε, σημειώνει τα πάντα. Έχουμε πολλή δουλειά λοιπόν ε, να κάνουμε στο μέλλον, αλλά αν μπορώ να προσθέσω μία πτυχή η οποία θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερο σημαντική, είναι και ο διακοινοβουλευτικό διάλογος. Γιατί το κοινοβούλιο έχει αντιπροσωπείες για διατλαντικέ σχέσει για την, σχέσεις με άλλες χώρες. Οπότε και σε αυτά τα θέματα ε, και αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να ε, ε, παρισφρήσουν στον δια... κοινοβουλευτικό διάλογο που κάνετε με τις τρίτες χώρες. Νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμο. Ευχαριστώ. ως Αμερικάνος που ζω εδώ και 7 χρόνια στην Ευρώπη και πραγματικά αγαπώ πολύ αυτή τη χώρα, την Ήπειρο, πρέπει να διατηρήσουμε το διάλογο με τις ΗΠΑ. Πείτε τους τι θέλετε η δική, της, η δική τους η διαδικασία είναι ότι έρχονται εδώ και κάνουν διαβουλεύσεις με τον ΝΑΤΟ, μιλούν με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πείτε τους λοιπόν όταν μιλάτε τι θέλετε. Για την, υπάρχει πρωτοβουλία για την ε, ε, για τον πυρηνικό αφοπλισμό, αλλά πρέπει να ακουστεί η φωνή σας. Επίσης, ε, ε, μιλήστε με τη Ρωσία. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά μιλήστε με τη Ρωσία και μην ξεχνάτε τρίτον την Ασία. Ακούω πολλέ προτάσεις που λένε, εντάξει, α τους απαγορεύσουμε α πούμε, ε, τώρα ακούω διάφορες ε, συζητήσεις ε, όταν, όταν, όταν η, Ιαπωνία θύμισε στις ΗΠΑ ότι το να υπάρχει πυρηνικός εξοπλισμός δεν, κάνει τον, δεν καθιστά τον κόσμο ένα πιο ασφαλές μέρος. Ακούστε λοιπόν την Ασία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τις Φιλιππίνες, την Ταϊβάν. Και η Ευρώπη μπορεί νομίζω να συμβάλλει στην παγκόσμια ασφάλεια, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν όλους που ήσασταν εδώ σήμερα. Σας προτείνω ένα σύντομο διάλειμμα 20 λεπτών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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE βουβαλίου του του

pardonnez-moi, de ce petit euh, aparté. Et euh, je voudrais, en notre nom à tous, euh, dire quel est notre plaisir d'accueillir. Γεια σας και πάλι. Ε, έχουμε μαζί μας ε, τον κύριο Πιέρα Ντελσό για μια ανταλλαγή απόψεων. Είναι αναπληρωτή Γενικό Διευθυντής από τη Γενική Διεύθυνση Grow τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συζητήσουμε τι πτυχέ τη διαστημικής πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια. θέλουμε να συζητήσουμε ε, τα θέματα που αποτελούν προτεραιότητα για την Επιτροπή μας ε, και στο πλαίσιο της δημιουργίας αυτής της νέας Γενικής Διεύθυνσης ε, Βιομηχανικής Πολιτικής Έρευνας και Διαστήματος είναι πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Εκ μέρους των συναδέλφων σας εκφράζω το ενδιαφέρον όλων μας για μια στενή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να έχουμε μία ε, καλή συνεργασία με μια ειδική σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι το οποίο επιθυμεί και η εκλεγήσα πρόεδρος ε, Ursula Φόντερ Λάιεν. Η Ευρώπη ε, έχει ένα διαστημικό τομέα παγκόσμιας κλάσης ε, και η βιομηχανία κατασκευής δορυφόρων είναι εξαιρετική με 33% της παγκόσμιας αγοράς. Ο τομέας του ε, διαστήματος εξελίσσεται ταχύτατα και αυξάνεται και ο ανταγωνισμός με νέους παράγοντες από την Ινδία, Βόρεια Κορέα, Κίνα κλπ κάτι το οποίο ανοίγει φιλοδοξίες, ανοίγει και δυνατότητες, ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις για την ασφάλεια για όλα τα κράτη-μέλη. Η Ευρώπη θα πρέπει μαζί να προσπαθήσει να ενισχύσει τη θέση του ηγέτη στο χώρο του διαστήματος και να χρησιμοποιήσει αυτή την πολιτική ως μέσο για την ανάπτυξη της στρατηγικής της αυτονομίας. Στις Ηνωμένε Πολιτείες η πρόσφατη δημιουργία μιας στρατιωτικής διοίκησης Spacecom για ένα μελλοντικό στρατό του μέλλοντος δείχνει ότι το διάστημα έχει πρωταρχική σημασία για την ασφάλεια και την άμυνα. Η υλοποίηση του διαστημικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021-2027 πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει παγκόσμιος ηγέτης και παράλληλα εποφελείται από τις δυνατότητες που προσφέρει ο χώρος του διαστήματος για την ασφάλεια της Ευρώπης, δημιουργώντας συνέργειες μεταξύ των διαφόρων τομέων της άμυνας και του μη στρατιωτικού τομέα. Τα στοιχεία ασφάλειας αυτού του προγράμματος που αποτελούν πρωτοβουλίες για τις τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρου, και για τις ε, κυβερνητικές επικοινωνίες, ε, το gov.com, καθώς και για την επιτήρηση στο διάστημα, το SSA, με πιλωτικά ε, προγράμματα, τα οποία υποστηρίζονται από το Κοινοβούλιο, έχουν προϋπολογισμό μόνο 500 εκατομμύρια ευρώ. Και σε διεθνέ επίπεδο, τα θέματα διακυβέρνησης, τα οποία συζητούνται σε πολυμερή βήματα για την εκμετάλλευση των πόρων του διαστήματο και για την διαχείριση της ε, κίνησης στο διάστημα δείχνουν τη σημασία που έχει το να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο όπου ε, η αναζήτηση πόρων πάντοτε ήταν αντικείμενο διαφωνιών μεταξύ των κρατών. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του κυρίου Ντελσό. Σας δίνουμε το λόγο για 15 λεπτά το πολύ και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Ναι, είναι καλό να υπάρχουν τακτές επαφές και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου για ένα τέτοιο θέμα που ενδιαφέρει όλους τους Ευρωπαίους και γενικότερα όλο τον κόσμο. Στην εισαγωγή σας κάνατε μια καλή σύνοψη όλων των διακυβευμάτων, των θεμάτων που υπάρχουν και θα πρέπει όλα αυτά να τα παρακολουθήσουμε και να σας πω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, έχουν αυτό το space command, αυτή την, το, το, διαστημικό σώμα. Ε, και αυτό γιατί. Ε, είναι κατανοητό τι γίνεται με την πολιτική για το διάστημα στην Ευρώπη. θέλουμε όχι μόνο να εκτοξεύουμε δορυφόρους, αλλά θέλουμε αυτοί οι δορυφόροι να μας παρέχουν ε, μια σειρά υπηρεσιών. Η οικονομία μας ήδη έχει αυξημένη εξάρτηση από τους ε, δορυφόρους και ε, αυτή η τάση θα αυξηθεί στο μέλλον. Οπότε θα εξαρτάται όπως σήμερα και στο μέλλον η οικονομία μας από τους δορυφόρους. Άρα θα πρέπει να τους προστατεύσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι λογικό. Επομένως, η ΥΠΑ ΕΕ, που είναι βασικός παίκτη στο διάστημα, να θέλουν να προστατεύσουν αυτά που έχουν στο διάστημα. Γιατί θα είναι τρομερές οι συνέπειες μιας επίθεσης. Οπότε, για να εστιάσουμε σε ό,τι γίνεται στην Ευρώπη. Και εσείς τα είπατε ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε κάνει. Γιατί πολλές φορές θεωρούμε ότι οι άλλοι τα κάνουν καλύτερα, ότι λειτουργούν αλλού καλύτερα τα πράγματα. Κι όμως κάναμε τόσα πολλά με τον Γαλιλαίο και τον Κοπέρνικο. Ε, όσα κάναμε ήταν εξαιρετικά αξιόλογα, είναι επιτυχίες αυτά για τον Ευρώπη και συνεργαστήκαμε και γι' αυτό πετύχαμε. Να, ένα παράδειγμα το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Δεν είμαι ειδικό για τον Γαλιλαίο, αλλά και ούτε εσείς, αλλά αυτή τη στιγμή ο Γαλιλαίος είναι το ευρωπαϊκό GPS. Και κάποια στιγμή θα υπάρξει κάτι που θα λέγεται ο Αμερικανικός ο Γαλιλαίος, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ ε, αξιόλογο σύστημα. Τώρα, για αυτό που σας ενδιαφέρει, το θέμα της ασφάλειας υπάρχει ε, μια σειρά υπηρεσιών ο Γαλλιός και μεταξύ των οποίων είναι και μια υπηρεσία ανοιχτή σε όλους το ότι μπορείτε να του χρησιμοποιήσετε ε, με, στο, το τηλέφωνο, το κινητό, στο αυτοκίνητο έχουμε τώρα ένα δις συσκευών που χρησιμοποιούν τον Γαλλίο και αυτή η τάση είναι αυξητική. Άρα σε λίγο θα μιλούμε για δύο δις. Επομένως είναι κάτι που ωφελεί όλους, αλλά είναι και άλλες υπηρεσίες του Γαλιλαίου. Υπάρχει κάτι που είναι λιγότερο γνωστό, αλλά αφορά την ασφάλεια. Search and Rescue. Έρευνα και διάσωση, δηλαδή ότι έχουμε γεωεντοπισμό αυτών που κάπου έχουν χαθεί. Και κυρίως στην θάλασσα. Και αυτό γίνεται με μια ακρίβεια πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο μέσο ή εργαλείο. Και σήμερα κιόλας. Κοιτάξτε το Twitter ή το δικό μας website και μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα, μια επίδειξη ε, του πόσο γρήγορα κάποιος που είναι χαμένος στη θάλασσα εντοπίζεται γιατί έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και άλλο ένα στοιχείο που είναι σημαντικό το PRS Public Related Services και αυτό είναι θέμα ε, που έχει σχέση με την ασφάλεια είναι μια υπηρεσία η οποία προστατεύει και αφορά κάποιους δέκτες που μπορούν να συνεργαστούν με αυτή την λειτουργία. Να σας εξηγήσω τι γίνεται. Εάν μπορεί να υπάρξει κάποια σύγκρουση κάπου στην Ευρώπη, ε, κάπου στον κόσμο, υπάρχει ένα ανοιχτό σήμα το οποίο μέσω Γαλιλαίου και GPS σας έρχεται. Ε, και αυτό τότε θα κοπεί Επομένως ε, δεν θα μπορείτε να ξέρετε που είστε σε αυτή την περίπτωση. Μόνο επομένως όσοι έχουν αυτούς τους δέκτες του PRS ε, με το κρυπτογραφημένο σήμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την υπηρεσία. Άρα σε περίπτωση σύγκρουσης ε, είναι πάρα πολύ βασικό να έχει κανείς αυτό το προστατευμένο σύστημα το οποίο όμως το έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι και βέβαια οι στρατιωτικοί γιατί εκείνοι θα πρέπει να έχουν την ευκολία του γεωεντοπισμού. Άρα το GPS, ο Γαλιλαίος μας λένε που είμαστε και που μπορούμε να πάμε. Άρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό η περίπτωση. Εδώ σταματάω για τον Γαλιλαίο και θα δούμε μετά τα υπόλοιπα. Υπάρχει και ο Κοπέρνικος. Είναι ένα σύστημα παρατήρησης της γης. Συνεχώς φωτογραφίζει την γη και δίνει μια σειρά υπηρεσιών πολύ χρησίμων για τη θάλασσα, για την ατμόσφαιρα, για την ε, μόλυνση, για την κίνηση ε, του εδάφους είναι και αυτό θέμα ε, ασφάλειας. Εάν, για παράδειγμα, έχουμε ε, μια πλημμύρα, έναν σεισμό, έναν ανεμοστρόβιλο μπορεί ο Κοπέρνικος πάρα πολύ γρήγορα να παράσχει τις φωτογραφίες και την περιγραφή ε, των σημείων που έχουν πληγεί από τα σχετικά φαινόμενα. Αυτό το ε, δίνουμε αυτή την υπηρεσία σε όποιους για να βοηθήσουν επί τόπου και επομένως είναι πιο εύκολος εντοπισμός. Δεν υπάρχει τίποτα σαν το Κοπέρνικο στον ε, κόσμο. Οπότε έχουν τέτοια φαινόμενα, ε, ανεμοστρόβιλους, ε, οι Αμερικανοί, ε, σεισμούς κλπ. Ε, έχουν και μας ζητούν τις υπηρεσίες του Κοπέρνικου. Άρα παρέχουμε τις υπηρεσίες στους Αμερικανούς διασώστες για να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Με τον Κοπέρνικο τώρα στο μέλλον τι θα κάνουμε. Εάν έχουμε την πρικοδότηση, εάν υπάρξει ο κανονισμός για το διάστημα, είναι το ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα ασφαλείας, δηλαδή παρατήρησης των συνόρων. Διότι και πάλι από το διάστημα μπορεί κανείς να τα δει όλα. Οπότε, εάν έχουμε τα χρήματα, θέλουμε αυτό να κάνουμε στο μέλλον, τέτοια υπηρεσία υποπτία συνόρων, θαλασσών ε, και όλο αυτό να είναι αποτελεσματικό για πολλές δουλειές. Δεν το έχουμε ακόμη αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλουμε να υπάρξει στο μέλλον. Και εάν φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα, θα υπάρξει ένα μικρό πρόβλημα. Πρέπει να λυθεί ότι το σύστημα αυτό για το οποίο σας μίλησα είναι ένα ανοιχτό σύστημα. Άρα όλες οι πληροφορίες θα είναι προσβάσιμες ε, από όλους. Αν θέλετε μπορείτε να δείτε όλα αυτά τα στοιχεία, όλες αυτές τις φωτογραφίες που είναι πάρα που πηγαίνετε στο Google Earth και θα τις δείτε. Οι περισσότερες φωτογραφίες του Google Earth είναι από τον Κοπέρνικο. Δεν το ξέρετε αλλά έτσι είναι. Αν θέλουμε μια κρυπτογραφημένη, προστατευμένη υπηρεσία για πιο συγκεκριμένα μέτρα, ε, τότε θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να μην ε, είναι γενικευμένη χρήση Οπότε αυτά. PRS για τον Γαλιλαίο και για τον Κοπέρνικο που ήδη χρησιμοποιείται για τα θέματα διάσωσης. Ε, όλα αυτά θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για ε, επιχειρήσεις επιτήρηση των συνόρων, αν υπάρχει το χρήμα τώρα. Για το διάστημα ακόμα δεν έχουμε τα σχετικά, δεν είναι η πρόοδος του προλογισμού. Θα κάνουμε τα εξή. Πρώτα-πρώτα θέλουμε Συγγνώμη, έχουμε όλα αυτά τα αρχικά στη διάλεκτό μας. Ε, υπηρεσίες ασφάλειας πρώτα-πρώτα μέσω δορυφόρου. Γιατί όταν υπάρχει κάποιο συμβάν, κάποιο περιστατικό, τότε οι υπηρεσίες εδάφους δεν ε, λειτουργούν. Πρόκειται για το GOVSAT. Κυβερνητική υπηρεσία, δηλαδή δορυφόρο. Οπότε δεν δουλεύουν υπηρεσίε εδάφου και αλλά χρησιμοποιούνται κάποια άλλα συστήματα τα οποία δεν είναι προστατευμένα, είναι ανοιχτά. Οπότε χρησιμοποιούμε τους δορυφόρους και έχουμε επομένως επικοινωνία τέτοια κρυπτογραφημένη μέσω του δορυφόρου. Και η διαφορά από τον Κοπέρνικο και τον Γαλιλαίο είναι η εξή στο Γαλιλαίο και στο Κοπέρνικο. Ε, εκεί εμείς έχουμε τους δορυφόρους και το πρόγραμμα. Τώρα στο gov.com όταν λειτουργήσει φαίνεται αλλιώς η κατάσταση. Κάποια, κάποια κρατημέλη, συγκεκριμένα κρατημέλη, θα έχουν την δυνατότητα αυτού του είδου της δορυφορικής ε, προστατευμένη και επικοινωνίας. Και αυτό που θέλει η Κομισιόν είναι να έχει αυτό το pooling and sharing, δηλαδή να χρησιμοποιείται αυτή η δυνατότητα που υπάρχει από κάποια κρατημέλη. Επίσης μπορούμε να αγοράσουμε από τον ιδιωτικό τομέα ε, κάποια εργαλεία και αυτά να τα δώσουμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Σε αυτού δηλαδή που δεν έχουν δορυφόρους, που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στου δορυφόρου και αυτοί να μπορούν να έχουν την πρόσβαση μέσω των δυνατοτήτων που δίνονται από τι μεγάλε χώρε. Οπότε χρησιμοποιούμε το ότι υπάρχει σε κάποια κράτη-μέλη και αυτά όλα τα δίνουμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό θέλουμε να φτιάξουμε και χρειαζόμαστε και τον ανάλογο προϋπολογισμό για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό και τον GovSat.com. Κάτι άλλο τώρα σημαντικό που και αυτό είναι στο σχέδιο κανονισμού είναι SST Space Surveillance Tracking είναι αυτά τα αρχικά SST δηλαδή έχουμε τους δορυφόρους στο διάστημα και καλά νομικός είμαι οπότε τι να πω και εγώ λέω ότι είναι ένας χώρος το διάστημα άδειος αλλά δεν είναι έτσι ναι είναι άδειο, αλλά έχουμε όλες αυτές τις ε, τροχίες που είναι γεμάτες από αντικείμενα, από πράγματα. Άρα ένα σωρό δορυφόροι, αλλά και πάρα πολλά σκουπίδια, στα πούμε, τα οποία είναι εκεί και βρίσκονται σε τροχιά. Ακόμα και ένα μικρό κομματάκι μπορεί να καταστρέψει έναν ε, δορυφόρο και αυτό έχει γίνει επανειλημμένα. Δηλαδή κάποιοι κάτι άγραστο, κάτι, ένα σκουπίδι να χαλάσει το δορυφόρο. Οπότε θα πρέπει να προσέχουμε τι γίνεται στο διάστημα, πού βρίσκονται αυτά τα απορρίμματα σε σχέση με τους δορυφόρους Αυτοί οι τόσο ακριβοί δορυφόροι θα μπορούσαν να χαλάσουν, να καταστραφούν και το πρόβλημά μας τώρα είναι ότι μόνο κάποια κράτη-μέλη έχουν τα απαραίτητα που τους επιτρέπουν να προσέχουν τι γίνεται στον ουρανό. Αλλά τα πιο πολλά τα έχουν οι Αμερικανοί. Οπότε εξαρτώμεθα σε αυτό το σημείο από τους Αμερικανούς για να μας δώσουν δηλαδή τις απαραίτητες πληροφορίες. Και βέβαια με τα ενδεχόμενα μειονεκτήματα που μπορεί να έχει αυτό. Ας πούμε πρόσφατα ενδεικτικά είχαμε έναν ευρωπαϊκό δορυφόρο σε τροχιά και την τελευταία στιγμή και ήρθε ένας άλλος δορυφόρος και μας είπαν οι Αμερικανοί ότι θα είναι στην ίδια τροχιά και θα πρέπει να το μετακινήσουμε. Άρα έπρεπε εμείς και οπότε όλα αυτά έγιναν για να μην έχουμε τη σύγκρουση με τον άλλο δορυφόρο που ήταν δορυφόρος του Elon Musk. Οπότε, να, όπως και στο GovSat.com Χρησιμοποιούμε αυτό που έχει κάποιο κράτος μέλος, χρηματοδοτούμε ούτω ώστε να αυξηθούν οι πόροι και όλες οι πληροφορίες που μαζεύονται από τα κράτη-μέλη παρέχονται σε όλους. Και έτσι να μην εξαρτώμεθα από τους Αμερικανούς. Το πρόβλημα είναι για να τα λέμε όλα είναι το εξής ότι εάν προσέχουμε όλα αυτά τα σκουπίδια και όλους τους δορυφόρους, τότε έχουμε και παρατήρηση και εποπτεία και των στρατιωτικών δορυφόρων, ε, το οποίο βέβαια δεν ενθουσιάζει και τόσο πολύ κάποια ότι δηλαδή τελικά οι πληροφορίες για τις κινήσεις των στρατιωτικών δορυφόρων είναι γνωστές σε όλους, οπότε βλέπουμε ότι θα πρέπει από τη μία να ξέρουμε τι γίνεται στο διάστημα, αλλά από την άλλη θα πρέπει να προστατεύουμε τους στρατιωτικούς δορυφόρους. Άρα αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα, δύσκολο πρόβλημα, δεν έχουμε ακόμα τη λύση του, άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να το εξετάζουμε. Οπότε φτάνω στο τελευταίο σημείο για το διάστημα και μετά θα δούμε για την άμυνα. Ε, για το διάστημα είναι κάτι άλλο, το οποίο είναι σημαντικό για το μέλλον. Και δεν λέω για μια δεκαετία ή δεκαπενταετία, λέω για κάτι το οποίο αφορά την διαχείριση της ε, κίνησης των ε, δορυφόρων, της κυκλοφορίας τους. Γιατί είναι βέβαια τεράστιο το διάστημα, αλλά οι τροχιές και ο χώρος των τροχιών είναι πραγματικά περιορισμένος. Οπότε, εκεί πραγματικά τα πράγματα είναι στριμωγμένα, περιορισμένα και ίσως θα ξέρετε ότι στις ΕΠΑ υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να εκτοξεύσουν ε, ε, κάποιους σχηματισμούς ε, δορυφόρων εκατοντάδων ή και χιλιάδων. Και ήδη όμως είναι πάρα πολύ σε τροχιά. Οπότε πώς κανείς μπορεί να εκτοξεύσει καινούριου. Και το θέμα το οποίο τώρα τίθεται είναι το πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση της πρόσβασης στο διάστημα. Και έχουμε ε, στο ΝΑΤΟ δουλειά και προχωρεί η δουλειά εκεί πέρα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι Αμερικανοί αποφάσισαν να προχωρήσουν μόνοι τους. Οπότε είπαν ε, εμείς θα αποφασίσουμε ε, πώς εσείς θα έχετε πρόσβαση στο διάστημα και έχουν επίσης αρχίσει να επεξεργάζονται το θέμα. Και εμείς το ίδιο. Τι θα κάνουμε άρα, αφήσουμε εκείνους να τα αποφασίσουν όλοι. Ε, βέβαια, υπάρχει και το, τονάτο που είναι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να υπάρξει διάλογος με τους Αμερικανούς, ούτως ώστε να έχουμε κοινού κανόνες και έτσι να μπορούμε να αποφασίσουμε από γενού τι γίνεται στο διάστημα. Και βέβαια και θέλουμε όπως και εσείς διαφάνεια, αλλά ε, δεν θέλουν όλα τα κράτη-μέλη το ίδιο, γιατί αν υπάρχει ε, ρύθμιση του διαστήματος, τι θα γίνει με τους έτοιμους δορυφόρους, τι θα κάνουμε. Άρα δεν το θέλουν τόσο διακαώς όλα τα κρατημέλη αυτό. Σας είπα πως έχει το τοπίο. Φαντάζομαι θα έχετε ερωτήσεις. Τώρα για να δούμε τι γίνεται με αυτό το Ταμείο Άμυνας. Πρώτα πρώτα αυτό το Ταμείο ε, κάθε αυτό δεν υπάρχει και ακόμα δεν υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ των συνομοθετών για αυτό το Ταμείο σας λέω για το ενδεχόμενο κείμενο το οποίο θα ισχύσει. Πρόκειται τώρα για ένα πρόγραμμα, ισχύει για δύο χρόνια, ε, η ADP ονομάζεται, στα αγγλικά δεν ξέρω στα γαλλικά, ε, ισχύει προσωρινά, το οποίο είναι πρόγραμμα ανάπτυξης της ε, αμυντικής βιομηχανίας. Δεν δούμε τώρα τι σχέση έχει το διάστημα με αυτά. Όπως και είπα στην εισήγησή μου, έχουμε ένα σωρό θέματα τα οποία έχουν σχέση με την άμυνα είπαμε το PRS για το Γαλιλαίο, το GovSatcom, σας είπα και το SST και αυτό το οποίο που σκεπτόμαστε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, δεν αποφασίζουμε εμείς μόνοι μας ως Κομισιόν, ε, τελικά όλα μαζί τα κράτη-μέλη με την υποστήριξη της Κομισιόν. Επομένως, στον τομέα της άμυνας είναι σαφές ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να θεωρήσουν ότι τους συμφέρει να κάνουν κάτι στην άμυνα μέσω του διαστήματος. Και εδώ έχουμε ένα σωρό προγράμματα τα οποία πρόκειται να ε, είναι επιλέξιμα για αυτό το ταμείο. Ποιε είναι οι προποθέσει, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρει επιχειρήσει τριών κρατών μελών που να συνυποβάλλουν ένα πρόγραμμα. Δεν μπαίνω στι λεπτομέρειε, ξέρω ότι είστε ειδικοί εδώ, αλλά δεν είναι θέμα το ότι η Κομισιόν δίνει κάποιους πόρους για να αναπτύξει ε, κάποιες δυνατότητες. Πρώτη για τεχνολογίες που αναπτύσσονται για κάποια προγράμματα που τα αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις με τη βοήθεια των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, η Κομισιόν για να βοηθήσει την τεχνολογία ε, συγχρηματοδοτεί. Οπότε έχουμε τέτοια προγράμματα, ιδίω όσον αφορά την εποπτεία, την παρατήρηση του SST, το GovSatcom, για τις ε, κυβερνήσεις, αλλά όσον αφορά αυτό το ταμείο στην τελική του μορφή, που ενδεχομένω αυτό είναι, θα γίνει το 21, είναι σαφές ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε τη διάσταση του ε, διαστήματος για να μπορέσουμε να έχουμε τη χρηματοδότηση των εθνικών προγραμμάτων. Γιατί είπαμε, δεν είναι ουδέτερο το διάστημα, δεν είναι ένα χώρο που πολλά είναι ρόδινα και αθώο, είναι πάρα πολύ σημαντικό οικονομικά και καθ' αυτό το διάστημα, αλλά και σε σχέση με όσα γίνονται στην γη. Οπότε γι' αυτό ε, η σχέση μεταξύ άμυνας, ταμείου και διαστήματος είναι κάτι που ένα και έχει μεγαλύτερη σημασία. Εδώ σταματώ γιατί ξύντλησα το χρόνο μου. Συγγνώμη που μακρηγόρησα και ευχαρίστω να απαντήσω τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι ήταν πάρα πολλά αυτά που μας είπατε γιατί είναι ένα θέμα που αξίζει να το συζητήσουμε διεξοδικά και μάλιστα στην παρούσα κατάσταση με όλα αυτά τα οποία γίνονται στην Ευρώπη. Μας μιλήσατε για τις φιλοδοξίες που μπορούμε να έχουμε για την επιτήρηση του διαστήματος, καθώς και για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, πριν να δώσω το λόγο στους συντονιστές, γιατί προτείνω να ζητήσουμε από κάποιους ομιλητές να κάνουν τις πρώτες ερωτήσεις και να απαντήσετε σε όλες μαζί. Σε θέματα επιτήρησης του διαστήματος, θα μπορούσαμε ε, να δούμε το βαθμό εξάρτησης της Ευρώπης από τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αν έχουμε μια φιλοδοξία αυτονομίας για την Ευρώπη, με όλες τις δυσκολίες και τους δισταγμούς που έχουμε, ποια πρέπει να είναι η πορεία που θα ακολουθήσουμε. Αγνώ Ντονζόν, εκ μέρους του Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Ντελσό για την παρουσίασή σας που ήταν ιδιαίτερα επεξηγηματική και πολύ έντιμη και ακριβής γιατί μας υπενθυμίσατε τα όρια που υπάρχουν και τα προβλήματα που συνεχίζουν να τίθενται. Μας υπενθυμίσατε ότι πολλά από αυτά που συζητάμε για το Ευρωπαϊκό Υπερταμείο ακόμη ε, είναι λίγο θεωρητικά. Ε, μπορεί να υπάρχει ενθουσιασμός στις πρωτεύουσες και καμιά φορά και προς τις τράπεζες, αλλά είναι πάρα πολλά αυτό που πρέπει να γίνουν, άρα πρέπει να είμαστε ακόμη σε επαγρύπνηση. Ένα σχόλιο μάλλον παρά ερώτηση είναι το εξής. Σήμερα όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θεωρούν το διάστημα, μιλώ τώρα για την άμυνα, θεωρούν το διάστημα ως ένα νέο χώρο πιθανών ε, συγκρούσεων. Στη Γαλλία και στην Ιταλία βλέπουμε να γίνονται σιγά σιγά παραγγελίες για το διάστημα εκ μέρους ε, των ε, ενόπλων δυνάμεων και οι εθνικές βιομηχανίες κινητοποιούνται για να έχουν κάποιο πάτημα στο διάστημα. Τα κονδύλια για τα οποία μιλάμε είναι πολύ μεγάλα. Καμία χώρα της Ευρώπης μόνη της δεν έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει επαρκείς πόρους για την πρόσβαση, την επιτήρηση και όλα αυτά τα οποία πάρα πολύ σωστά μας περιγράψατε. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μια παράδοξη λοιπόν διτή κίνηση. Από τη μια πλευρά κατανοούμε ότι πρέπει κάποια πράγματα να κινητοποιήσουμε για να έχουμε δυνατότητες. Από την άλλη πλευρά όμως Υπάρχει, υπάρχουν οι εθνικοί ανταγωνισμοί που ξεκινάνε μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών και χρειάζεται χρόνος για να τα συγκεντρώσουμε όλα. Έχουμε χάσει χρόνο. Ε, και εγώ θα ήμουν υπέρ του να έχουμε ένα ευρωπαϊκό υπερταμείο το οποίο θα επενδύσει μεγάλα ποσά στο διάστημα. Υπάρχουν άλλοι τομείς στου οποίους ξέρουμε να συνεργαζόμαστε για τους χερσαίου εξοπλισμούς, ακόμη και για την πολεμική αεροπορία. Ήδη ξέρουμε να συνεργαζόμαστε, ήδη έχουμε βιομηχανίε που έχουν τη δυνατότητα, που έχουν τα χρήματα. Εδώ τώρα μιλάμε για νέα πράγματα που ανοίγονται για το διάστημα. Αυτό ήταν το σχολείο μου. Ευχαριστώ, κύριε Ζουιβιέχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Γενική Διευθυντά για την παρουσίαση. Ήταν πάρα πολύ καλή. Και τα σχόλια της Πρόεδρου ήταν επίσης πολύ εύστοχα. Σχετικά με τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως είπατε, το 1 τρίτο των δορυφόρων κατασκευάζονται στην Ευρώπη, το 60% στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην Ευρώπη και στρατιωτική και μη στρατιωτική. Αναφέρεται το πρόγραμμα Γαλιλαίος. Στο μέλλον, μέσα από συνεργασίες θα φτάσουμε. Και ο διαστημικός χώρος είναι ένας χώρος για τον οποίο είναι απαραίτητη η συνεργασία. Αναφέρεται το Γαλιλαίο που είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο πολλές χώρες είναι υπερήφανες, είμαστε όλοι υπερήφανοι γι' αυτό. Υπάρχει αντίστοιχα το GPS. Ποιο είναι το κόστος για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνεργασία. Ε, δώστε μας μια τάξη μεγέθους για τα κονδύλια που απαιτούνται. Κάτι άλλο τώρα για την στρατιωτικοποίηση του διαστήματος. Έχουμε μια συνθήκη του 1967, μια συνθήκη που έρχεται από μια άλλη εποχή. Είχαμε τη δυτική πλευρά και το σοβιετικό μπλοκ από την άλλη. Και μιλούσαμε για την απόρριψη των όπλων μαζικής καταστροφής. Για το 1967 οι προοπτικές ήταν διαφορετικές. ο αφοπλισμός των δορυφόρων επικοινωνίας μπορεί να αποτελέσει όπλο μαζικής καταστροφής σήμερα. Είναι διαφορετικές οι έννοιες που συζητάμε. Ποια είναι η προσέγγιση μας λοιπόν έναντι της συνθήκης του 1967. Αρνούμεθα την στρατιωτικοποίηση του διαστήματος, αλλά σε τι βαθμό και ποια είναι η συλλογική μας προσέγγιση και τι μέσα προτείνεται για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Πέτρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον κύριο Ντουσό καταρχάς. Έχω ένα ερώτημα για το Κοπέρνικους. και το πρόβλημα του ελέγχου των ευρωπαϊκών συνόρων. Είπατε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό στο μέλλον, όχι προς το παρόν, αλλά χρειαζόμαστε προπολογισμό. Τι προϋπολογισμό δηλαδή χρειάζεστε για να υπάρξει έλεγχος των ε, ευρωπαϊκών συνόρων. Και δεύτερον, υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας. Και τρίτον, είπατε ότι ίσως να υπάρξει πρόβλημα με την επικοινωνία, γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια όταν ε, ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρον είναι όταν κάνουμε τη συζήτηση για τη Frontex και τον έλεγχο των συνόρων, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο συνολικό θέμα της μετανάστευσης. Είναι λοιπόν ένα σημείο αρκετά ενδιαφέρον που θα μπορούσαμε, στο οποίο θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε, γιατί ξέρω ότι χρειάζονται πάνω από 10.000 αξιωματούχοι για να ελέγχουν τα σύνορα, οπότε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Η τεχνολογία τι μπορεί να κάνει. Οι δορυφόροι βλέπουν τα πάντα. Άρα αυτό είναι το ερώτημά μου. Επικοινωνία, Προπολογισμό χρονικός ορίζοντας. Και πώς θεωρείτε εσείς ότι μπορεί ο Κοπέρνικος να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση των συνόρων. Ευχαριστώ. Merci. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριο Μίξα. Ε, Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Δεν θα πω ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τα τεχνικά του θέματος του διαστήματος και των τεχνολογιών και των δορυφόρων, αλλά πριν από λίγες μέρες, μάλιστα χτες, το συζητήσαμε εδώ στην Επιτροπή, το θέμα των α, επιθέσεων the, στα στενά του Ορμούς. Και στη συζήτηση αυτή υπόθηκε ότι υπάρχουν συστήματα είτε εξαρτημένα είτε αυτόνομα που χρησιμοποιούνται και από τους συμμάχους μας και από τους εχθρούς μας, θα μπορούσα να πω. Με διαχείριση από μακριά για την πλοήγηση κτλ. Σίγουρα υπάρχει μεγάλο δυναμικό και ευκαιρίες ώστε αυτές οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες και σε εμπορικούς δηλαδή πάροχους υπηρεσιών, αλλά βεβαίως αυτό προφανώς έχει αρκετούς ε, κινδύνους. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση την επίθεση ήταν ένα σύστημα που διαχειριζόταν μέσω. Ε, είχαν διαχείριση δορυφορική για την επίθεση. Αλλά το ερώτημά μου είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να μετριάσουμε λιγάκι αυτού του κινδύνου για να μπορούν αυτές οι υπηρεσίες να χρησιμοποιηθούν και από εμπορικούς ε, εμπλεκόμενους φορείς. Και μάλιστα για τη συζήτηση που κάναμε το πρωί για την ε, μη πυρηνική διάδοση και τις διάφορες συνθήκες. Ένας από τους ομιλητές μας προειδοποίησε να μην ξεχνούμε την Ασία. Μήπως μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό. Μιλούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ συχνά και τον ανταγωνισμό που υπάρχει και τη συνεργασία που ίσως υπάρξει. Η οπτική από την πλευρά της Ασίας ποια είναι, η της Κίνας, της Ινδίας κυρίως, για τέτοιου είδους συστήματα πλοήγησης και χρήσης των τεχνολογιών διαστήματος. Merci, Christophe Ευχαριστώ, Christophe Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, μιλήσατε και για το PRS. Οι κρυπτογραφημένες επικοινωνίες θα έχουν στρατηγικό ρόλο στο μέλλον. Με την υπόθεση Snowden είδαμε ότι η παρακολούθηση θυνόντων από το NSA δεν ήταν κάτι που χαροποίησε την Ευρώπη και με το σύστημα PRS θα υπάρχουν λύσεις αλλά από ό,τι έχω ακούσει ζήτησαν πρόσβαση στο σύστημα PRS οι Ηνωμένε Πολιτείε, στο ευρωπαϊκό σύστημα PRS. Μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε αυτό. Όντως ζήτησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε πρόσβαση στην τεχνολογία μας. Για την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος, το SST. Τώρα μπορεί να έχουμε 2.000 ε, δορυφόρους, στο μέλλον μπορεί να έχουμε τεράστιο αριθμό. Στην Επιτροπή Ήτρεχτες ε, μας αναφέρεται ότι έχετε κάποιες ανησυχίες για τον προϋπολογισμό που δίνουμε στο διάστημα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις στη σημερινή Επιτροπή που είναι ασφάλειας και άμυνας τι είδους ανησυχίες είναι αυτές που τρέφεται και αν κινητοποιήσουμε ένα τέτοιο υπερταμείο, παράλληλα θα κινητοποιήσουμε και ιδιωτικούς πόρους για να έχουμε κάποιες λύσεις για την πολιτική του διαστήματος. Στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, δεν ανησυχούν για την SpaceX ή αντίστοιχες πρωτοβουλίες, γιατί έχουν τεράστια κονδύλια. Εσείς έχετε πραγματική ανησυχία για τη χρηματοδότηση της διαστημικής πολιτικής ή θα καταφέρουμε να βρούμε λύσεις. Κύριε Γενική Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις. Ξεκινώ με την πρώτη σας ερώτηση. Ε, σε ποια μέτρα εξαρτώμαστε από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Όντω ορισμενα ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ε, δυνατότητες, ε, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα ιδιάζον καθεστώ αυτή τη στιγμή και η Ισπανία έχει επίση κάποιε δυνατότητε. Κυρίω όμω οι δυνατότητες προέρχονται από τι Ηνωμένε Πολιτείε, δηλαδή αυτή τη στιγμή η πληροφόρηση έρχεται από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Μα δίνουν πληροφορίε όταν θέλουν και ό,τι πληροφορίε θέλουν να μα δώσουν. Παραδείγματο χάρη, δεν πάει πολύ καιρό που ένα κινέζικο δορυφόρο έπεσε που θα μπορούσε να έχει πέσει οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη. Μας είπαν οι Αμερικανικές αρχές ότι θα πέσει ο δορυφόρος κάπου ανάμεσα στη Βόρειο Θάλασσα και στη Σιβηρία. Δεν μας έδωσαν λοιπόν και ακριβέστατες πληροφορίες. Τελικά έπεσε ο κινέζικος δορυφόρος σε ένα σημείο που δεν ενόχλησε κανέναν, αλλά εξαρτώμεθα από τους Αμερικανούς απολύτως για την πληροφόρηση που μας δίνουν. Έχουμε υπογράψει μια συμφωνία με τα πέντε κράτη-μέλη που σας ανέφερα για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες για την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος, προσπαθώντας να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη ενημέρωση. Στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες επενδύσεις από περισσότερες χώρες και να έχουμε ένα είδος συγκέντρωσης των πόρων. Το ερώτημα του κ. Ντανζόν για το ε, ε, Ταμείο Άμυνας ε, ε, υπάρχει πρόταση, αλλά κανείς δεν έχει υπογράψει την επιταγή και δεν μπορώ εγώ να υπογράψω την επιταγή. Στον τομέα του διαστήματος και στον τομέα της άμυνας έχουμε την εντύπωση ότι επειδή έγινε η πρόταση από την Επιτροπή, υλοποιήθηκε κιόλα. Κάθε άλλο, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και γι' αυτό απευθύνομαι σε εσά, τους Ευρωβουλευτές, για να εξηγήσετε και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι το διάστημα και η άμυνα είναι ιδιαίτερα σημαντικοί τομείς για όλους τους λόγους που προαναφέραμε και είναι πολύ ουσιαστικό το να υπάρχει καλός προϋπολογισμός. 13 δισεκατομμύρια για την άμυνα δεν είναι τίποτα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και είναι εντελώς ε, μηδαμινό σε σχέση με το τι δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. 16 δις που προτάθηκε για την, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι τίποτα σε σχέση με το τι έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι όμως απαραίτητο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Κύριε Ντανζό, πολύ σωστά είπατε ότι βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι συνειδητοποιούμε ότι το διάστημα είναι ένα διακύβευμα και γι' αυτό χρειάζεται προστασία των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν μπορεί το κάθε κράτος μόνο του να κάνει κάτι, γιατί υπάρχει και η στρατιωτική διάσταση, αλλά και οικονομικά, αν δεν πιστούν όλοι ότι πρέπει να συγκεντρώσουμε τους πόρους, δεν θα καταφέρουμε τίποτα επειδή υπάρχουν δυνατότητες σε κρατικό επίπεδο, μια απότομη προσέγγιση της Επιτροπής που θα τα συγκέντρωνε όλα δεν θα είχε θετικά αποτελέσματα. Χρειάζεται λοιπόν με ένα σωστό με σωστό παιδαγωγικά τρόπο να πείσουμε όλους ότι πρέπει να συμφωνήσουν και χρειάζεται χρόνος και είναι και πολύπλοκο, αλλά είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε. Το Ταμείο Άμυνας που ελπίζω ότι θα τεθεί σε λειτουργία, ελπίζω σύντομα, αν μπορέσει να μας δώσει δυνατότητες για ανάπτυξη τεχνολογιών και για διαστημική τεχνολογία θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εσείς ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη-μέλη μπορείτε να περάσετε το μήνυμα αυτό στα κράτη-μέλη. Για την ερώτηση του κυρίου Ριβιέρ, αυτό που είπατε για τη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος, ε, όντως το κείμενο υπάρχει και δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτά που είναι ήδη γραμμένα. Τώρα βέβαια τα διακυβεύματα είναι διαφορετικά γιατί μπορείτε με λέιζερ να καταστρέψετε δορυφόρους. Υπάρχουν τεχνολογίες. Οι κίνδυνοι τους οποίους αντιμετωπίζουμε τώρα είναι διαφορετικής μορφής. Δεν είναι η πυρηνική βόμβα που φοβόμαστε για το διάστημα, αλλά μπορεί οι ακτίνες λέιζερ να διακόψουν τις δορυφορικές ε, επικοινωνίες και μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες σε εκατομμύρια πολίτες αυτό. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πώς θα προστατεύουμε ε, τα μέσα που έχουμε στο διάστημα. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν θα πετάξουμε αυτά τα οποία έχουμε ήδη από το παρελθόν, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα στο μέλλον, γνωρίζοντας ότι τώρα είμαστε σε ένα νέο πλαίσιο, σε ένα νέο περιβάλλον. Ο Κοπέρνικο ε, τώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατεύσουμε τα σύνορα, για τον απλό λόγο ότι αν θέλει κανεί να προστατεύσει τα σύνορα, εντάξει, μπορούμε να τα φωτογραφίσουμε. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό είναι πολύ μεγάλο ο χρόνο. Οπότε, αν δει κανεί ε, κάτι σε μια συγκεκριμένη φωτογραφία σε ένα μέρο, δεν φτάνει σε αυτό το μέρο τόσο γρήγορα για να δει τι γίνεται. Οπότε, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο τρόπο που θα είναι πολύ πιο ακριβές, ε, που θα είναι πολύ πιο ακριβής ο τρόπος αυτός και πολύ πολύ συγκεκριμένος. Στη νέα πρόταση ε, Έχουμε τρία, τρεις διαφορετικές αποστολές που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Μία είναι η, ε, παρακολούθηση του α, ε, του άνθρακα για, για το περιβάλλον, για τα αέρια του θερμοκηπίου κτλ. Δεύτερον, πάλι σχετίζεται με το α, ε, περιβάλλον, είναι η παρακολούθηση του, των αρκτικών, για την, πάλι για, το, για την προσοχή του περιβάλλοντος. Και τρίτη αποστολή μας, η παρακολούθηση των συνόρων. Η παρακολούθηση των συνόρων τώρα. Έχουμε κάνει κάποιου υπολογισμού, ξέρουμε πώ θα κοστίσει. Δεν θα κοστίσει τόσο πολύ. Εντάξει, βέβαια για μένα είναι πολλά λεφτά, αλλά είναι λιγότερο από 2 δισευρώ. ευρώ. Το ερώτημα βέβαια είναι ότι αν δεν έχουμε ε, χρήματα για να διατηρήσουμε τον Κοπέρνικο, τι κάνουμε. Αν δεν έχουμε χρήματα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Θα επικεντρωθούμε στην παρακολούθηση του ε, του άνθρακα, των αρκτικών ή των συνόρων. Αυτή την συνάντηση θα πρέπει να την πάρουμε μαζί με τα κρατημέλη, βέβαια. Δεν θα είναι εύκολο, σίγουρα. Το καλύτερο σενάριο θα ήταν να έχουμε αρκετά κονδύλια για να μπορούμε να καλύψουμε και τι τρει αποστολέ. Σε σχέση τώρα με το χρονικό ορίζοντα, ε, με το, για το διάστημα πρέπει να, να κατανοήσει κανείς ότι ε, χρειάζονται πολλά χρόνια από τη στιγμή που παίρνει κάποιο μια απόφαση μέχρι να την πραγματοποιήσει τελικά. Οι, οι δορυφόροι δεν λειτουργούν ε, μέσα σε μέρες, αλλά αν δεν πάρουμε μια απόφαση δεν θα φτάσουμε ποτέ στο στόχο μας. Και το θέμα της ασφάλειας τώρα, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στο τρέχον πλαίσιο όλες οι πληροφορίες είναι δημόσιες που έρχονται για το Κοπέρνικο. Αλλά όταν μιλάμε για τα σύνορα και τη διαχείριση, προφανώ δεν μπορούμε να είναι δημόσιε αυτέ οι πληροφορίε. Οπότε πρέπει να βρούμε μια διαφορετική δίωδο επικοινωνία για να έχουν τι πληροφορίε μόνο αυτοί που τι χρειάζονται. Η Frontex, τα κρατημέλη. Και στο ΣΑΤΣΕΝ είχαμε πει ότι θα μπορεί να αναλάβει τέτοιου είδου ε, δραστηριότητε. Οπότε ε, για την ασφάλεια πρέπει να έχουμε διαφορετική δίωδο επικοινωνία. Ε, συγγνώμη τώρα που πάω από το ένα θέμα στο άλλο για την ερώτηση του κυρίου Γκουτλέ για το PRS και για την πρόσβαση των Αμερικανών. Ε, πρέπει να κατανοήσετε ότι το σύστημα PRS, όπως σας είπα, δυνητικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση σύγκρουσης, σε περίπτωση στρατιωτικής έντασης. Γιατί έχει αναπτύξει η Ευρώπη τον Γαλιλαίο, διότι το GPS είναι ένα στρατιωτικό σύστημα που δόθηκε σε μη στρατιωτικές χρήσεις, αλλά εξαρτάται από τους Αμερικανού Αμερικανούς στρατιωτικούς. Και η Ευρώπη είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση όπου εξαρτώμεθα από τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί στη ΣΥΠΑ και γι' αυτό αναπτύξαμε τον Γαλιλαίο. Τώρα, το σύστημα PRS που ακόμη είναι υπό εξέλιξη, δεν έχει τελειοποιηθεί, είναι ένα σύστημα που θα δίνει αυτές τις κρυπτογραφημένες πληροφορίες. Αυτό που συζητάμε τώρα με τους Αμερικανούς είναι το εξή, γιατί όντως κάνουμε συζητήσεις με τους Αμερικανούς και τους Νορβηγούς, αυτό είναι γνωστό. Και για, την, ε, ε, ε, για το Brexit επίσης συζητούνται παρόμοια θέματα. Δεν θα δώσουμε πρόσβαση στους Αμερικανούς για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται το σήμα. Οι συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή αφορούν το τι θα γίνει σε περίπτωση προβλήματος. Εάν το στρατιωτικό σύστημα GPS δεν λειτουργεί, μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί δείκτες που θα τους δίνουν το σήμα PRS. Δηλαδή, να σας πω ποιος είναι ο φόβος, ότι αν υπάρχει μια σοβαρή επίθεση κατά του Αμερικανικού συστήματος GPS, το στρατιωτικό σύστημα GPS, δεν θα έχουν πλέον σύστημα γεωεντοπισμού. και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα PRS. Δηλαδή δεν αναπτύσσουμε το σύστημα PRS μαζί με τους Αμερικανούς, ούτε τους δίνουμε πρόσβαση και έλεγχο του PRS, αλλά μπορεί να τους δώσουμε πρόσβαση στο σήμα σε περίπτωση προβλήματος. Αυτό συζητάμε τώρα με τους Αμερικανούς και τους Νορβηγούς και ίσως να ενδιαφέρει και άλλες χώρες στον κόσμο. Δεν θα το δώσουμε στους Κινέζους βέβαια, αλλά αυτή είναι η λογική. Για τον προϋπολογισμό αυτό που είπα είναι ότι υπάρχουν προτάσεις για τον προϋπολογισμό αλλά ακόμη έχουμε πολλά να υλοποιήσουμε. Για τη χρήση των δορυφόρων, κύριε Μίξερ, είναι ξεκάθαρο ότι το διάστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αρνητικά. Το σήμα που έρχεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για drones κλπ. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ένα, μια πτυχή του Γαλιλαίου που την ονομάζουμε ταυτοποίηση δεν είναι το PRS, δεν είναι οι υπηρεσίε για το κοινό. Συγγνώμη που τα λέω έτσι λίγο μπερδεμένα. Ε, και εγώ δεν είμαι τεχνικό από ε, αυτών των θεμάτων και προσπαθώ να τα πω όπω τα έχω καταλάβει. Τι σημαίνει, ότι θα υπάρχει ένα τρόπο σύντομα να στείλει κανεί σήμα σε όλου που θα εγγυάται ότι το σήμα αυτό έρχεται από το Γαλιλαίο. Τι θα πει αυτό συγκεκριμένα. Α πούμε ότι μια μέρα έχουμε ένα αυτόνομο αυτοκίνητο και του λέτε θέλω να με πας στο σπίτι. Βάζει την ε, διεύθυνσή σου ή τέλο πάντων είναι το δικό σου αυτοκίνητο, ξέρετε τη διεύθυνσή σα. Οπότε, αν κάποιος παρέμβει, με το, παρέμβει στο σήμα που έρχεται από το GPS, θεωρείτε εσεί ότι σας πηγαίνει το αυτοκίνητό σας σπίτι, αλλά το αυτοκίνητο θα σας πάει αλλού, κάπου που δεν θέλετε. Με το Γαλιλαίο θα έχουμε ένα σήμα όπου θα μπορεί κανείς να είναι σίγουρος ότι το σήμα που έρχεται δεν έρχεται από κάποιον άλλον, έρχεται όντως από το σύστημα Γαλιλαίο. Οπότε θα λέτε στο αυτοκίνητο θέλω να πάω σπίτι και θα είσαστε σίγουρος ότι ο Γαλιλαίο θα σας πάει σπίτι σας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το GPS δεν την έχει αυτή τη ε, δυνατότητα, τη λειτουργία. Και αυτό είναι κάτι για, πολλές, για πολλές ε, εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δεν είναι το PRS, είναι κάτι άλλο. Και τελευταίο σημείο. Μίλησα για τη ΣΥΠΑ. Η Κίνα όμως είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Η Κίνα ε, επενδύει μαζικά στο διάστημα. Έχουν ε, εκτοξεύσει ε, χιλιάδες δορυφόρους, έχουν βάλει πάρα, πολλούς, πάρα πολλούς πόρους για το διάστημα. Οπότε αυτό ήδη είναι μια ένδειξη του ότι θεωρούν ότι είναι στρατηγικό στοιχείο το διάστημα και επενδύουν σε αυτό δεν δαπανούν τα χρήματα έτσι απλώς για να κάνουν την επένδυση. Ε, βάζουν πραγματικά κόπο και χρόνο και χρήμα για να γίνει η επένδυση. Οπότε ναι, είπαμε, αλλά η Κίνα είναι η πιο μεγάλη μας ε, πρόκληση για το, για το διάστημα. Έχουν εμπορικού, φυσιολογικού, έχουν ε, κανονικού αλλά και στρατιωτικού δορυφόρου. Οπότε. Και όπως είπατε κύριε Γκρουντλέρ, πρέπει να εξασφαλίσουμε δημόσιε επενδύσει. και για την άμυνα και για το διάστημα, γιατί συνδέονται. Χρειάζονται λοιπόν δημόσιε επενδύσει, αλλά χρειάζονται και ιδιωτικέ επενδύσει. Θέλουμε οι ιδιώτε επενδυτέ να έρθουν και να επενδύσουν. Χρειαζόμαστε όλου του ε, τομεί πρέπει να ανοίξουν. Είναι πολύ σημαντικοί οι παίκτε, έχουμε πολύ καλέ εταιρείε ε, πρώτη γραμμή, υψηλή ποιότητα. Πρέπει να επενδύσουν και να φέρουν και νέα σκεπτικό, νέε νοοτροπίε για το πώς μπορεί κανείς να δουλέψει στο διάστημα. Αλλά αυτό δεν θα το αποφασίσω εγώ. Αυτή όμω είναι μία από τι βασικέ ε, προκλήσει που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τον νέο κανονισμό για το EDF και για το διάστημα. Και σίγουρα χρειάζονται περισσότερε ε, ε, επενδύσει στον τομέα αυτό. Συγγνώμη και πάλι μακρηγόρησα. Καθόλου. Δίνω το λόγο στον Μίχαλ Γκάλερ που είχε μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ένα θέμα που δεν αναφέρεται αλλά που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι κάνουμε γενικές συζητήσεις για τη στρατηγική αυτονομία στον τομέα της άμυνας και όσον αφορά το διάστημα υπάρχει η έννοια της ε, τεχνολογικής μη εξάρτησης. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω αν η νέα σας γενική διεύθυνση θα ασχοληθεί και με το θέμα αυτό. Είναι θέμα της συζήτησης για τη στρατηγική αυτονομία. η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία είναι πολύ σημαντική. Βασικά το θέμα είναι αν θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτονομία για την Ευρώπη σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, να μην εξαρτώμεθα από τεχνολογίες που προέρχονται από αλλού. Εσείς είστε ειδικό για το θέμα, αλλά το λέω και για άλλους που μπορεί να μην είναι ειδικοί. Γι' αυτό το διευκρινίζω. Αν μιλάμε για ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας στο διάστημα και στην άμυνα, πρέπει να δημιουργήσουμε ανεξαρτησία. Αν μιλάμε για το διάστημα, τώρα που συζητάμε τον Γαλιλαίο, η διάσταση ασφάλειας του Γκαλιλαίου είναι ότι θέλουμε να το αναπτύξουμε με ευρωπαϊκές τεχνολογίες. Θέλουμε στην Ευρώπη να αναπτυχθούν τεχνολογίες. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε ήσυχοι ότι σε στρατιωτικές σειράξεις θα χρησιμοποιήσουμε τον Γκαλιλαίο, δεν θα το επηρεάσει κάποιος μη Ευρωπαίος. Και στο πλαίσιο του Brexit είναι και αυτό μία από τις συζητήσεις που γίνονται, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη του Γκαλιλαίου και του PRS όταν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, εάν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί δεν θέλω να συζητήσουμε για τον Brexit, δεν θα είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στο PRS. Για την άμυνα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, την ίδια προσέγγιση ακολουθεί. Θέλουμε να αναπτύξουμε τεχνολογίες που θα είναι σημαντικές για την Ευρώπη και θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να έχουν τις τεχνολογίες που θέλουν. Κάτι που είναι σημαντικό για την άμυνα ε, είναι ότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι πολλά κράτη-μέλη είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Το θέμα των τεχνολογιών λοιπόν είναι ότι δεν θα πρέπει να είναι και σε αντίφαση με Τη τεχνολογία του ΝΑΤΟ και η νέα εκλεγήσα πρόεδρος της Επιτροπής ε, σαφώς ανέφερε ότι υπάρχει η σχέση μας με το ΝΑΤΟ και θα πρέπει να αποφύγουμε τις ε, συγκρούσεις. Δεν θα είμαστε απολύτως ανεξάρτητοι από ολόκληρο τον κόσμο, αλλά θα αναπτύσσουμε τις δυνατότητες που θέλουμε στην Ευρώπη, έχοντας κατά νου το γενικότερο πλαίσιο. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει η νέα Γενική Διεύθυνση, γιατί δεν είναι ακόμη εδρεωμένη. Θα έχουμε νέο επίτροπο, δεν θέλω να προδικάσω για τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Οπότε προς το παρόν αυτά μπορώ να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, όχι, κανείς μας δεν θεώρησε ότι μακρηγορήσατε γιατί ενδιαφερόμαστε και θέλουμε να συνεχιστεί η συζήτηση για το θέμα. Αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε τι κάνει η υπηρεσία σας ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε το κεκτημένο που υπάρχει, Μα είπατε τι γίνεται με τον ε, Γαλιλαίο, τον Κοπέρνικο, την αυτονομία στο διάστημα και όλα αυτά τα οποία σήμερα αποτελούν ε, κίνδυνο για αυτές μας τις ε, υποδομές, για τις επιχειρήσεις, για τον κόσμο. Εάν δεν μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους δορυφόρους μας και τις σχετικές υποδομές. Ευχαριστούμε για την ανταλλαγή απόψεων. Ε, πέρα στις συνεδριάσεως και θα τα ξαναπούμε στις 8 Οκτωβρίου.